Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Αναφορών. Στο σημείο 2, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Σας ζητώ να σημειώσετε την αναβολή του σημείου 9 κατόπιν ετήσεως του κυρίου Μαριά θα εξετάσουμε αυτή την αναφορά στις 30 Μαΐου. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Έχω κάποιες ανακοινώσεις. Από τη συνεδρίαση των συντονιστών που ολοκληρώθηκε μόλις πριν πείτε στην αίθουσα, λάβαμε τις εξής αποφάσεις, αιτήματα για, από τις ομάδες για τις κατοπινές ημερήσιες διάταξης. Προσωρινή ημερήσια διάταξη του Ιουνίου εγκρίθηκε με κάποιες μικρές τροποποιήσεις η αναφορά για την υψηλή τάση συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη για... του Ιουλίου ακριβώς για εκθέσεις και γνωδοτήσεις. Λαμβάνουμε γνώση της επιστολής ε, του Προέδρου της Επιτροπής Απασχόλησης προς εμένα και θα συνεχίσω τις διαπραγματεύσεις μαζί του για να πετύχουμε την ενεργοποίηση του άρθρου 54. Εφόσον δεν γίνει θα το ξανασυζητήσουμε. Αιτήματα για αναφορές αυτά που σας είπα και για τα σημεία Β, η αναφορά 248 και 242 και 692 παραμένουν ανοιχτές. Η 248 έκλεισε μάλλον, οι άλλες δύο παραμένουν ανοιχτές. για τις διερευνητικές επισκέψεις και αποστολές. Καταγράφουμε το σχέδιο προγράμματος για τον Τάραντα στην Ιταλία. Είναι μια επίσκεψη που θα ξανασχεδιάσουμε τώρα γιατί αναβλήθηκε στο παρελθόν και η γραμματεία έχει λάβει εντολή να αλλάξει κάπως τη σειρά των ε, συναντήσεων, να τροποποιηθεί το πρόγραμμα. Οι συντονιστές ενέκριναν το σχέδιο προγράμματος για την ακρόαση στις 22 Ιουνίου για την ανάκτηση της εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα και αποφασίσαμε να εγκρίνουμε το πρόγραμμα με κάποιες αλλαγές. Θα επανέλθουμε με τη γραπτή διαδικασία. Οι συντονιστές επίσης ενέκριναν το προσωρινό πρόγραμμα για τους απάτριτες και αποφάσισαν να προσκαλέσουν εμπειρογνώμονες όπως πρότειναν το ΕΛΚ και οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Στην διερευνητική επίσκεψη στην Ισπανία 22 και 23 Μαΐου το πρόγραμμα ε, εγκρίθηκε. Και επίσης συμφωνήσαμε να ζητήσουμε γραπτές συνεισφορές από τις περιφερειακές αρχές που εμπλέκονται στο όλο θέμα στην Ισπανία, ώστε να έχετε κάτι να διαβάσετε κατά την πτήση. Για την αναφορά Αντωνιάννα, Συμφωνήσαμε να συμπεριλάβουμε την πρόταση για αποστολή διερευνητική στον κατάλογο των ενδεχόμενων διερευνητικών αποστολών για το πρώτο εξάμεινο το 2018 και αυτό το αποφασίσουμε τον Οκτώβριο φέτος. Έχουμε λοιπόν ένα μακροσκελέστατο κατάλογο και θα δούμε τι θα επιλεγεί. Οι συντονιστές έλαβαν γνώση των ε, προ σημείων και δεν υπήρξε κάτι επιπλέον στα διάφορα όπως ανακοινώθηκε και προηγουμένω. Ναι, Βεβαίω ενημέρωσα του συντονιστέ ότι μία πρόταση για πιλωτικό, έχουμε λάβει μία αίτηση για πιλωτικό πρόγραμμα και θα υποβληθεί στην Επιτροπή Προπολογισμών για μία πρώτερη αξιολόγηση. Επίση ενημέρωσα του συντονιστέ για τη σημερινή ανταλλαγή απόψεων που είχα το πρωί με έναν δικαστή, μάλλον ένα μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου. Αυτά τώρα μπορούμε να τα αφήσουμε και να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ελπίζω ότι ήδη έχετε δοκιμάσει τις κάρτες σας, τα μηχανήματα, αν λειτουργούν. Και από τα χαμόγελά σας βλέπω ότι έτσι είναι. Ρομπέρτα, έχεις κάρτα? Α, έρχεται. Ωραία. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μία κυρία που θα ανέβει με το χέρι και θα ψηφίζει έτσι. Ψηφίζουμε λοιπόν για το ομάδα εργασία για τα θέματα παιδική πρόνοιας. Κάποιο ζητά το λόγο. Σολεδάδ, παρακαλώ. Να πω απλώς ότι δεν έχω κάρτα για την ώρα. Οπότε παρακαλώ να μα μετρήσετε και εμά. Ωραία. Είναι λοιπόν η ισοπαλία έτσι, γιατί έχουμε έναν από το ΕΛΚ και έναν από του Σοσιαλιστέ και δημοκράτε χωρί κάρτα. Εξισορρόπηση να περάσουμε στην ψηφοφορία για την σύσταση αυτή. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Έχει αποσυρθεί 4. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να κάνουμε έλεγχο. Έξι, Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Φυσικά και δεν δουλεύει αφού δεν έχετε κάρτα. Α, έχετε κάρτα. Πέρας της ψηφοφορίας. είναι ένας υπεράριθμος από το ΕΛΚ. Είπαμε το χέρι, όχι και κάρτα, Ρόμπερτα. Εντάξει, κάποιο μπορεί να βγάλει την κάρτα του, έτσι, συμφωνείτε. Να επαναλάβουμε την ψηφοφορία, επαναλαμβάνουμε. Άρχεται η ψηφοφορία, επαλήθευση για την τροπολογία 6. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 8. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9 και 10. Ταυτόσιμες. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 11. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12. Υπέρ, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 και 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αυτή να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Με πολλές, πολλές αποχές. 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ. Α, καταπίπτει δεν εγκρίθηκε, απορρίφθηκε. Νομίζω ότι καλά τα λέω. 21 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μετά κατά τμήμα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 31 και 32 από κοινού υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά αποχές πρέπει να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται, απορρίπτεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να κάνουμε έλεγχο. 39. Άρχεται ψηφοφορία για έλεγχο. Πέρας. Εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 42 υπέρ, Κατά. Αποχές. Να κάνουμε έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία για την 42. Πέρας. Απορρίφθηκε. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Πρώτο τμήμα. Πρώτο τμήμα, πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, αγκρίνεται Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έλεγχος. Έλεγχο. Επαλήθευση. Οκ. Okay. Άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα. Πέρας. Απορρίφθηκε. 47 και 48 από κοινού. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 53 και 54 από κοινού. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 55 υπέρ, κατά, να κάνουμε έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία για την 55. Πέρας. Από... Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58 και 59 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τελική ψηφοφορία. ηλεκτρονική αυτή. Πέρας. ένα επιπλέον κατά από κάποιον που δεν έχει δικαίωμα ψήφου. 17 υπέρ, 13 κατά. Εγκρίνεται. Και έτσι ολοκληρώνουμε τις σημερινές μας ψηφοφορίες. Κυρία Πιτέρα, έχετε το λόγο. Παρακαλώ, ακούστε την κυρία Πιτέρα. Πρόεδρε, λυπούμε εκ μέρους του ΕΛΚ, λυπούμε που αναγκαστήκαμε να καταψηφίσουμε έτσι όπως διαμορφώθηκε το κείμενο, διότι αρχικά είμαστε υπέρ για την σύσταση της ειδική ομάδας. Η ομάδα συστάθηκε μετά από πρωτοβουλία του ΕΛΚ μάλιστα, και περιμέναμε διακαώς τα πορίσματα 18 μηνών εργασίας, ώστε να μεταφραστούν και σε πρακτικές συστάσεις και δράσεις. Δυστυχώς οι συστάσεις αυτές βασίστηκαν σε μονόπλευρη προσέγγιση και προκειμένου να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των γονέων και όχι τόσο των παιδιών Δεν είχαμε μάλιστα καμία θετική εξέταση σχετικών αναφορών από όσε λάβαμε σε αυτό το διάστημα. Είναι ακόμη ανοιχτέ. Δεν περατώθηκε η εξέτασή του. Δεν είμαστε λοιπόν ικανοποιημένοι με τα πορίσματα και γι' αυτό δεν είχαμε άλλη επιλογή παρά να καταψηφίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για αυτές τις διευκρινήσεις, ε, ε, για την πολιτική σας τοποθέτηση ως ΕΛΚ. Πέτερ. Ναι. Να πω απλώς ότι είχαμε υποβάλει μια πρόταση αποκινούμε την ομάδα Άλντε και θα ήθελα αυτό να καταγραφεί στα πρακτικά παρόλο που δεν ψηφίστηκε η προπολογία. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μια ψηφία ένα έγγραφο, μια τοποθέτηση που εξηγεί τη δική σας θέση στα πράγματα. Ολοκληρώνεται η συζήτηση περί της ψηφοφορίας σήμερα. Να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε με τη σημερινή ημερήσια διάταξη και φτάνουμε στην αναφορά 1233 για τις κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά. Παρουσία του αναφέροντος. Σας παρακαλώ όσοι έχετε σκοπό να φύγετε από την αίθουσα, να το κάνετε ησύχω, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα. So, Mrs. Estrella... Κυρία Εστρέλα Γκόμες Βίνιας, η αναφέρουσα είστε μαζί μας. Θα σας δώσω το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, ένα στα τέσσερα κορίτσια και ένα στα έξι αγόρια την χάνουν κακοποίηση στην παιδική του ηλικία. Ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των παιδιών δέχονται τη βία αυτή εντό τη οικογένειά του η συγχρονική κακοποίηση και οι περιπτώσεις αιμομιξίας είναι αυτές ε, οι περιπτώσεις που δημιουργούν μεγαλύτερα ποσοστά. Είναι δύσκολο να βρεθεί δικαιοσύνη για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011-92 ε, δεν έχει μεταφερθεί επαρκώς στην Ισπανική νομοθεσία. Και αυτό σημαίνει ότι ε, η μαρτυρία του θύματος εξακολουθεί ε, να γίνεται με έναν τρόπο αρκετά αδιαφανή. Δεν υπάρχει προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες και στις ανάγκες του θύματος. Έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο αυτό στα παιδιά και είναι μη αποτελεσματική η διαδικασία. Δεν υπάρχουν απαρκή μέτρα προστασίας καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Και ποινικά και αστικά. Ξεκινάμε με το τεκμήριο ότι το θύμα δεν έχει δίκιο. Ερχόμαστε εδώ για να ε, επιβεβαιώσουμε κάποια πράγματα. Δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να μπορέσει κάποιος ε, να ε, επιβεβαιώσει την, ε, το κατά πόσο η ιστορία που λέει ένα παιδί είναι αληθινή ή όχι. Επειδή ένα παιδί ξαφνικά την ώρα που μιλάει κρύβει το κεφάλι του ή κρύβεται, θεωρείται ότι λέει ψέματα. Πολλά παιδιά λοιπόν δεν έγιναν πιστευτά στα δικαστήρια. Μιλάμε λοιπόν για διάκριση και λόγω φύλου και λόγω ηλικία. Υπάρχει ε, διάκριση λόγω ηλικία, διότι λέμε ότι ένα νέο, ε, ένα δικαστή λέει α πούμε ότι ένας, ένα παιδί δεν θέλει να δει τον πατέρα του, τότε θα πρέπει να έρθει στα συγκαλά του. Επίσης, άλλοι δικαστές λένε ότι συχνά τα παιδιά λένε πράγματα που δεν έχουν νόημα. Ε, τα παιδιά όντω δυσκολεύονται να γίνουν πιστευτά από το δικαστικό σύστημα. Είναι διάκριση λοιπόν αυτή. Το δικαίωμα στο, που έχει το, το θύμα να μπορέσει να ανακτήσει την αξιοπρέπειά του σημαίνει ότι θα πρέπει να το δεχτούν και οι δύο γονεί του. Ακόμα και αν ο ένα από του δύο είναι ε, ε, κατηγορούμενος. Όταν ε, η, μητέρα είναι αυτή που κατηγορεί και ο κατηγορούμενος είναι ο, ο πατέρας, τότε δεν ισχύουν οι ίδιοι κανόνες. Παίρνονται αποφάσεις για νέους και για παιδιά, αγόρια και κορίτσια, αυθερέτως. Υπάρχει συχνά απόρριψη από το παιδί προ τον δράστη, ο οποίο συχνά είναι μέρο τη οικογένειά του, και αυτό δεν γίνεται αποδεκτό από το δικαστήριο. Δεν μπορούμε να σα δώσουμε βέβαια στοιχεία γι' αυτό, διότι δεν υπάρχει κάποιο επίσημο όργανο το οποίο να συλλέγει ε, τέτοιου είδου στοιχεία. Στον φάκελο που έχει συμπεριληφθεί στο αίτημα έχουμε βεβαίω εκθέσει που αξιολογούν και καταδεικνύουν τα κενά στο δικαστικό σύστημα. Υπάρχει το σύνδρομο τη απομάκρυνσης από του γονεί. Ε, τα δικαστήρια δεν λαμβάνουν υπόψη αυτά. Εδώ έχουμε μια σειρά από περιπτώσεις όπου βλέπουμε όλα αυτά τα, στα οποία αναφερθήκαμε. Ε, καλό θα ήταν βεβαίω να πούμε ότι πολλέ μητέρε δεν θέλουν να συνεργαστούν λόγω φόβου. Ζητούμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει από το, από το κράτο τη Ισπανία να βελτιώσει το ισπανικό σύστημα είναι, πρέπει να είναι σαφές ότι να είναι συγκεκριμένες προθεσμίες παρέμβασης. Θα πρέπει να, να υπάρξει προσαρμογή στις ανάγκες του κάθε αγοριού και κοριτσιού. Να υπάρχουν συγκεκριμένα τεχνολογικά δεδομένα και στον χώρο που λαμβάνει η χώρα η δίκη και στους χώρους αναμονής και βεβαίως να υπάρχει απόλυτη προστασία καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Θα πρέπει να πάρθουν τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να μην μπορεί πια να εφαρμοστεί αυτό το σύνδρομο ε, από του ως βάση για να μην γίνει δεκτή η μαρτυρία του παιδιού ή για να παρθούν μέτρα σε αστικό επίπεδο. Θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση της πρόσβασης των θυμάτων στη ψυχολογική αρρωγή ακόμα και αν δεν συμφωνεί ο κηδεμόνας, ο οποίος είναι κατηγορούμενος στην προκειμένη περίπτωση. Ε, αυτό που έχει σημασία είναι να λάβει η χώρα μια πραγματική σε βάθος αλλαγή στο πώς προσεγγίζει κανείς σε δικαστικό επίπεδο αυτής της περιπτώσης κακοποίηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την απάντηση. Κυρία Κάθριν Μπάουερ Μπούλστ είναι η εκπρόσωπος τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για σήμερα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως θα θυμάστε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, απέστειλε τις παρατηρήσεις της για την αναφορά αυτή από τον Οκτώβριο φέτος. Βάσει τη συμβολής της αναφέρουσας είχαμε εντοπίσει τρεις τομείς ενδεχόμενης παραβίασης ε, της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 93 του 2011. Πρώτα απ' όλα για την συγκεκριμένη διατύπωση του ισπανικού άρθρου που καλύπτει την υποχρέωση να ε, προστατεύονται τα παιδιά σε ποινικέ έρευνες και διαδικασίες η οδηγία προβλέπει ότι τέτοια προστασία θα προσφέρεται, αλλά το πρωτογενές δίκαιο εξαρκεί. Ε, αυτό βεβαίως μπορεί να προκαλέσει ενδεχομένως κάποιες ε, ε, διαφωνίες Πρώτα απ' όλα στην προστασία για το καλύτερο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, όπω ανέφερα και αναφέρουσα, και επίση την έλλειψη επιμέλεια στι δικαστικέ διαδικασίε και τι έρευνε, τι ανακρίσει. Συγκεκριμένα την έλλειψη προστασία του παιδιού κατά τη διάρκεια των διαδικασιών. Όπω ε, ενημερώσαμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να δώσει συνέχεια στην ε, διερεύνηση του θέματο. Έχουμε συμφωνήσει τώρα τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε και θα αποστείλουμε επιστολή προ τι Ισπανικέ Αρχέ την ερχόμενη εβδομάδα για να ζητήσουμε περισσότερε πληροφορίε για αυτού του ενδεχόμενου ε, τομεί παραβίαση τι οδηγίε. Ευχαρίστω να απαντήσω σε οτιδήποτε επιπλέον ερωτήσει μπορεί να έχετε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για αυτήν την σαφή τοποθέτηση και τώρα ο λόγος ε, στους συναδέλφους. Η κυρία Βαλίνα πρώτη. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω ε, τις ενώσεις που βρίσκονται πίσω από αυτήν την αναφορά και να τη συγχαρώ ε, διότι πραγματικά με αυτή την αναφορά μας εξηγούν τις επιπτώσεις μιας νομοθεσίας που οδηγούν σε καταστάσεις όπου ανήλικοι δεν έχουν την απαραίτητη προστασία. Οι υποψίες αυτών των ενώσεων που υποστηρίζουν ε, αυτήν την αναφορά είναι εξαιρετικά βάσιμες είναι λοιπόν ε, πολύ πιθανό η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία αυτή τη στιγμή να μην εφαρμόζεται σωστά, το είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώ και η οδηγία περί δικαιωμάτων των θυμάτων. Επίση γίνεται αναφορά ότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα στα δικαστήριά μα, ε, όπω ε, συγκεκριμένη επαγγελματική αντιμετώπιση των θυμάτων, στέγασή του. Ε, και υπάρχει πιθανότητα η χάρτη θεμελιών δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωσης να παραβιάζεται. Παραβιάζεται διότι έχει σχέση με τι σχετικέ οδηγίε. Έτσι λοιπόν συμφωνώ απόλυτα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι απαραίτητο να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Θα πρέπει να αναλύσουμε πολύ προσεκτικά τις πληροφορίες που θα ζητήσουμε και θα μας δώσουν οι Ισπανικές Αρχές και στη συνέχεια ε, θα πρέπει να περιμένουμε την έκθεση της ε, Επιτροπής και να λάβουμε όλες τις απαραίτητες εξηγήσει. Και για μια φορά συμφωνούμε με αυτό που απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πολύ ευαίσθητο το ζήτημα αυτό, πολύ λεπτό και ανεξάρτητα από τις πολιτικές μας προτιμήσεις πρέπει όλοι να κάνουμε μια προσπάθεια για να επιληθούν τέτοιου είδου ζητήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να διευκρινίσω ότι θα δώσω τώρα το λόγο για να έχουν χρόνο τα μέλη της Επιτροπής πρώτα να πάρουν το λόγο και μετά σε συναδέλφους που δεν είναι μέλη αυτής της Επιτροπής, αν δεν έχετε αντίρρηση. Πολύ ωραία. Παρακαλώ, Ρώσα. Ναι, ε, συμφωνώ με αυτό που είπε η Άγγελα. Όντως, από ό,τι φαίνεται ε, και μετά από αυτά που είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η μεταφορά των, των ευρωπαϊκών οδηγιών ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την οδηγία ε, για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και το άρθρο 20 αυτής της οδηγίας είναι πολύ ε, νερωμένη στην Ισπανία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την προστασία των συμφερόντων του ανήλικου. Τώρα, για την οδηγία σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων, το εξετάζουμε ακόμα, ε, το θέμα της μεταφοράς. Ε, πάντως είναι προφανές ότι θα πρέπει να μην ανοιχτεί αυτή η αναφορά. Ε, θα πρέπει να δούμε αυτό, αυτός ο διάβολος επικοινωνίας, ε, η επιστολή που θα ε, αποσταλεί στις ισπανικές αρχές, να δούμε πού θα οδηγήσει, τι απαντήσεις θα λάβουμε, εάν δηλαδή η μεταφορά του άρθρου από τον 18 και 20 δεν έγινε με τον κατάλληλο τρόπο και κατά πόσο υπάρχει λοιπόν ένα κενό ε, ε επί της ε, του οποίου έχει απόλυτο δίκιο ο αναφερόμενος, αναφέρον μάλλον το να κάνει αυτή την αναφορά. Και βεβαίω πρέπει να γίνουν και απαραίτητε διορθώσει με βάση τι πληροφορίε που θα μα δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σολεδάδο. Ναι, ευχαριστώ Σεσίλια. Ε, δεν έχουμε μεγάλες διαφωνίε εδώ μετά από αυτά που είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σε σχέση με τους ανήλικους για ένα θέμα τόσο ευαίσθητο όπως το θέμα της κακοποίησης, της σεξουαλικής κακοποίηση. Θέλω να ευχαριστήσω ε, τους αναφέροντες ε, διότι αυτή η αναφορά έχει να δώσει φωνή τελικά σε αυτά τα παιδιά που συχνά δεν λαμβάνεται υπόψη ε, και δεν ε, υπάρχει επαρκής προάσπιση των συμφερόντων τους. Ε, χαίρομαι επίσης για την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά προφανώς και θα πρέπει να υπάρξει μια παρακολούθηση και να λάβουν χώρα οι απαραίτητε τροποποιήσει στην νομοθεσία για να μπορέσει να θωρακιστεί το συμφέρον των ανηλίκων. Ευχαριστώ κυρία Τανόκα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να στραφώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ενημέρωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διερευνήσει περαιτέρω το θέμα για να δει αν υπήρξαν παραβιάσεις συστηματικά. Εξ όσων κατάλαβα από την παρουσίαση της αναφέρουσας, προφανώς και είναι συστηματικές παραβιάσεις. διότι έχει γίνει κακή υλοποίηση της οδηγίας. Η ερώτηση μου λοιπόν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κατά πόσον δεν ξέρετε πώς θα το ε, χειριστείτε το θέμα ε, και πώς θα το διαμορφώσετε και για αυτό τα λέτε αυτά, διότι πρέπει να πούμε στις Ισπανικές αρχές πώς τις κρίνουμε αυτές τις παραβιάσεις. Δεν είναι μεμονωμένες υποθέσεις από ό,τι φαίνεται, είναι συστηματικές παραβιάσεις λόγω της ε, πλημελούς υλοποίηση υλοποίησης της οδηγίας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ για το λόγο. Φαίνεται να υπάρχει συμφωνία μεταξύ ημών και το ΕΛΚ το βλέπει το θέμα ως πολύ σοβαρό και ευαίσθητο. Υποστηρίζουμε τη θέση της αναφέρουσας ε, στηρίζουμε και την προσπάθεια και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καλωσορίζουμε τον μελλοντικό διάλογο με τις Ισπανικές Αρχές. Από την πλευρά του ΕΛΚ πιστεύουμε ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αναφορά για να συνεχιστεί η εξέταση του θέματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κυρία Αλβιόλ και μετά η κυρία Σέντρα Ροντρίγκε. Και μετά ολοκληρώνουμε τον κατάλογο των αγορητών οπότε θα ξανατοποθετηθεί η αναφέρουσα. Ευχαριστώ Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την αναφέρουσα ε, για το έργο της και για το γεγονός ότι έφερε αυτή την αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου λέει ότι ενδεχομένω να μην υπάρχει συμμόρφωση σε ό,τι αφορά την οδηγία με την εξολογική και τη εξολογικοποίηση αλλά και την προστασία των ε, θυμάτων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την, πρόσταση, την έλλειψη προστασία καθ' όλη τη διάρκεια τη διαδικασία των ανηλίκων και την έλλειψη ε, γρήγορη αντίδραση. Αυτό που θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να επιταχύνει κάπως τη διαδικασία. Τι εννοώ. Αυτή η αναφορά υποβάλλεται το 2015. Έχουμε φτάσει στο 2017 και ακόμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι έχει ξεκινήσει τη διαδικασία να ζητήσει πληροφορίες από τις αρχές. Ε, νομίζω ότι το θέμα αυτό είναι αρκετά σοβαρό έτσι ώστε η διαδικασία αυτή να επιταχυνθεί κάπως. Εγώ θα ζητούσα και στα πλαίσια της Επιτροπής Αναφορών να μην περιμένουμε αυτές τις διαδικασίες που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που καλά κάνει και τις διενεργεί αλλά εμείς ως Επιτροπή Αναφορών να συνοδεύσουμε αυτή τη διαδικασία, να απευθυνθούμε και εμείς και να εκφράσουμε την ανησυχία μας στις Ισπανικές Αρχές. Αυτό νομίζω ότι θα έρθει να ενισχύσει το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νομίζω ότι με κάποιο τρόπο αυτό θα μπορούσε να επιταχύνει την όλη διαδικασία. Διότι, επαναλαμβάνω, η αναφορά έχει υποβληθεί το 2015, μπορεί να υπάρχει μη συμμόρφωση με την οδηγία, όπω λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, οπότε νομίζω δεν θα ήταν καθόλου περιττό και εμεί ω Επιτροπή Αναφορών να κάνουμε κάτι και να μην περιμένουμε απλά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τουλάχιστον να εκφράσουμε την ανησυχία μα στι πανικέ αρχέ. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να βοηθήσει ώστε τα πράγματα να πάνε κάπω πιο γρήγορα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σέντρα Ροντρίγκεθ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να εκφράσω την απόλυτη υποστήριξή μου στις προτάσεις που υπέβαλε η αναφέρουσα. Επίσης ε, να ζητήσω η αναφορά να παραμείνει ανοιχτή. Ε, βεβαίως θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία της συζήτησης αυτής για να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτήν εδώ την Επιτροπή Αναφορών να εμβαθύνουμε κάπως ε, το ζήτημα και να εξετάσουμε γενικότερα πώς εφαρμόζονται όλες οι νομοθεσίες ευρωπαϊκές ό,τι αφορά την ισότητα, ό,τι αφορά την βία, ε, την ενδοοικογενειακή και ό,τι αφορά την κακοποίηση σεξουαλική. Διότι φτάνουμε συχνά σε αυτές τις καταστάσεις επειδή χρησιμοποιούμε ε, τελικά μια φαλοκρατική προσέγγιση ό,τι αφορά την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας. Και ήθελα να, να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτήν την ε, αναφορά που, σε αυτό το αίτημα που θα υποβάλλεται προς τις ισπανικές αρχές ε, σκοπεύετε να εξετάσετε και αυτό το σύνδρομο της απομάκρυνσης από τους γονείς που είναι κάτι που χρησιμοποιείται όπως λέγεται και στην αναφορά από την ισπανική δικαιοσύνη ε, και πώς θα εξετάσετε αυτό το θέμα ότι πρέπει να υπάρχει προσωπικό που να είναι καταρτισμένο για να μπορέσει να βοηθήσει να συνδράμει τα θύματα. Αυτά ευχαριστώ. Ναι, νομίζω ότι ήταν τόσο σαφή η απάντηση της Κομισιόν. Ε, ξέρουμε πολύ καλά τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Ε, οπότε να δώσω τώρα το λόγο στην αναφέρουσα, στην κυρία Γκόμες Βίνιας, για δύο ακόμα λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μας ε, για την απάντηση από αυτή την Επιτροπή αυτής της Επιτροπής. Ε, για μας ως συλλογικότητες που ασχολούμαστε με αυτά τα πολύ λεπτά ζητήματα είναι σημαντικό να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή να βρούμε έναν τρόπο έτσι ώστε να τεθεί επιτάπητος στο ζήτημα αυτό και να γίνει μια έρευνα για το τελικά τι κάνει η Ισπανική δικαιοσύνη με τις υποθέσεις αυτές. Είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα διότι είναι περίπλοκες αυτές οι καταστάσεις όπου ζουν τα παιδιά αυτά και οι οικογένειές τους ε, μας ρωτούσαν οι εμπλεκόμενοι μας ρωτούσαν τα θύματα αυτά μπορεί να συμβεί κάτι με αυτήν την διαδικασία εμείς δεν ξέρουμε τι να τους πούμε ακριβώς πρέπει λοιπόν να κινηθούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα ευχαριστώ ευχαριστώ σας ευχαριστώ και για το θάρρος που επιδείξατε και για την ε, δέσμευσή σας, ε, να αυταπάρνησή για την προσπάθεια αυτή. Βεβαίως ε, θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Θα πρέπει η Κομισιόν να συνεχίσει το έργο της. Θα μείνουμε ε, βεβαίως ανοιχτή γραμμή με τις Ισπανικές Αρχές. Θα επισταλεί και μια επιστολή σύντομα προς τις Ισπανικές Αρχές και νομίζω ότι μπορούμε να κινηθούμε παράλληλα. Μπορούμε να στείλουμε και μια επιστολή στην Ισπανική κυβέρνηση και εμείς, όπου θα εκφράζουμε την ανησυχία μας ε, για τις ε, ενδεχόμενες παραβιάσεις αυτών των δύο οδηγιών. Ε, ήταν σαφές νομίζω αυτό που ακούσαμε, έτσι ώστε να γίνει κατανοητό ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται έτσι ώστε να επιληθούν τα ζητήματα αυτά το συντομότερο δυνατόν και να γίνει μια σωστή μεταφορά της οδηγίας στην Ισπανία. Βλέπω ότι γνέφουν καταφατικά εδώ οι συμμετέχοντες. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε όλοι. Όλους σας ευχαριστούμε που ήρθατε μέχρι εδώ στις ε, αλλά και για την ε, συνεχή προσπάθειά σας και καλή επιστροφή. Περνάμε λοιπόν στην επόμενη αναφορά, την 2654 του 2014 έχει να κάνει με νομικό ζήτημα και ε, την αναφορά για τις δικαστικές δαπάνες 10 καθώς 2012. Ο αναφέρον είναι εδώ, ο κύριος Φρανσίσκο Βερντούν Πέρες. Θα του δώσω το λόγο για 5 λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας μεταφέρω το πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα αυτό των δικαστικών εξόδων σε ό,τι αφορά την προστασία των ευρωπαϊκών, των καταναλωτών αυτή η σημασία συνοψίζεται ε, σε ένα μόνο στοιχείο. Η νομοθεσία και η ευρωπαϊκή αλλά και η ισπανική την προστασία των καταναλωτών αυτή τη στιγμή αλλοιώνεται όταν ο καταναλωτή που απευθύνεται στο δικαστήριο για να μπορέσει να γίνουν αυτά τα δικαιώματά του αντιμετωπίζει δικαστικά έξοδα, δικαστικά τέλη που δεν του επιτρέπουν να έχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Δεν του επιτρέπουν να προσφύγει. Είναι πολλά τα ζητήματα, ο καταναλωτής πρώτα απ' όλα βρίσκεται σε μια μενεκτική θέση σε σχέση με τον επαγγελματία. Ε, επίσης, ε, ε όταν προσφέρει ένα καταναλωτή, αυτό είναι προ όφελο τη κοινότητα, όχι μόνο προ όφελο του ιδίου, το σύνολο τη κοινωνία Είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις που φτάνουν στο δικαστήριο, λόγω του κόστους. Και αυτό ε, έχει ως αποτέλεσμα να μην βρίσκουν το δίκαιο τους οι καταναλωτές. Είναι πολλά τα ζητήματα και πρέπει να πούμε ότι για να φτάσουμε σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας ενιαίο για όλου του Ευρωπαίου καταναλωτές, είναι απαραίτητο να υπάρξει μια εναρμονισμένη νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να μην επιτρέπει να απαιτούνται ε, τέλη έξοδα για τον καταναλωτή που θέλει να προσφύγει για να προσπίσει τα δικαιώματά του οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω λοιπόν να ζητήσω από αυτή την Επιτροπή, την Επιτροπή Αναφορών, προ όφελο όλων των καταναλωτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αφενό να μείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και αφετέρου να ξεκινήσει η απαραίτητη διαδικασία έτσι ώστε σε ένα προσεχέ μέλλον να εγκριθεί μια τέτοια νομοθεσία εναρμόνιση. Ζητώ, με βάση αυτό που το 216.2 του κανονισμού του, του Κοινοβουλίου να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία, μια ε, έκθεση πρωτοβουλίας μάλλον και να υποβληθεί μια πρόταση ψηφίσματος στο, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου με θέμα αυτό. Θα ήθελα να αναφερθώ εν συντομία στο έναυσμα αυτής της αναφοράς. Πρόκειται για μια καταναλώτρια η οποία ζητάει να ε, ένα συμβόλαιο που έχει να κάνει με τον νόμο 10 του 2012 έπρεπε όμως να πληρώσει 300 ευρώ μόνο για να ξεκινήσει τη διαδικασία. Το μισό δηλαδή του ελάχιστου μισθού στη χώρα μας. Ήταν πραγματικά δυσανάλογο το ποσό αυτό και παράνομο στην πραγματικότητα, διότι ουσιαστικά πρόκειται για περιορισμό δυσανάλογο του δικαιώματος ε, προσφυγής στο δικαστήριο με βάση και την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μετά από τέσσερα χρόνια διαδικασίας ούτε ένα δικαστήριο δεν μπόρεσε ε, να αξιολογήσει ότι είναι δυσανάλογο αυτό, δυσανάλογη αυτή η δαπάνη. Ω δικηγόρο εδώ και χρόνια πρέπει να σα πω ότι τα εθνικά δικαστήρια πολλέ φορέ δεν ακολουθούν την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ούτε την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και πρέπει, μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι ο εθνικό νομοθέτη, όποια πολιτική προτίμηση και να έχουν, ε, συχνά, όπως με την νομοθεσία 10-2012, δεν λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες στον τομέα των καταναλωτών. Ο νόμος 10 του 2012 έχει αναθεωρηθεί το 2015. Δεν υπάρχουν πλέον οι δαπάνες για τα φυσικά πρόσωπα, αλλά πρόσφατα το, το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ισπανίας είπε ότι θα τροποποιήσει ε, εκ νέου την νομοθεσία και είναι αβέβαιο, αβέβαιη η συνέχεια. Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης τι γίνεται στα άλλα κράτη-μέλη. Μέσω της διεκτικής πύλης e-justice της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο κόστος το δικαστικό, ε, με βάση τι πληροφορίε που έχει δώσει το κάθε κράτος μέλο σε ό,τι αφορά τι δαπάνε, έχουμε διαπιστώσει δύο στοιχεία. Πρώτον, υπάρχουν πολύ μεγάλε διαφορέ, πολύ μεγάλε αποκλήσει ό,τι αφορά αυτήν τη δικαστική δαπάνη από τη μία χώρα στην άλλη. Αυτό οδηγεί σε πολύ σημαντικέ διακρίσει, διότι κάποιοι Ευρωπαίοι καταναλωτέ πληρώνουν πολύ περισσότερο από ότι άλλοι για να προστατευτούν τα δικαιώματά του. Επιπλέον, έχουμε διαπιστώσει ότι στι πληροφορίε αυτέ για τι δαπάνε δεν γίνεται πουθενά αναφορά Στι δαπάνε στον τομέα τη προστασία του καταναλωτή. Δηλαδή τα κράτη-μέλη δεν λαμβάνουν υπόψη τι ιδιαιτερότητε τη προστασία του καταναλωτή όταν καθορίζουν αυτό το, το σύστημα δικαστικών δαπανών. Τελειώνοντα να πω ότι ο μόνο τρόπο για να φτάσουμε σε ένα ενιαίο και υψηλό επίπεδο προστασία των καταναλωτών είναι να υπάρχει μια νομοθεσία εναρμονισμένη που να καταργεί τι δικαστικέ δαπάνε για όλου του καταναλωτέ που θέλουν να βρουν το δίκιο του. Ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ερικ και είναι ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Ε, θα σας ακούμε στα σουηδικά αν θέλετε. Θα το ευχαριστηθώ ιδιαίτερος. Δεν θα χρειαστώ ακουστικά. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω τα σουηδογγλικά μου αν θέλετε. Έχετε λάβει απάντηση, την έχετε μπροστά Αυτό που λέμε στην απάντηση είναι ότι έγινε μια μελέτη μεταξύ άλλων για το κόστος των ε, δικαστικών δαπανών. Η μελέτη είναι σχεδόν έτοιμη. Έχω ένα προσχέδιο μαζί μου, ε, αφορά μια έκθεση για την Ισπανία και έχουμε μια καλύτερη εικόνα του τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά το κόστος και την ε, αναλογία σε σχέση με το βασικό μισθό, αυτό έχουμε να πούμε πως είναι εθνική αρμοδιότητα. Ο καθορισμός του κόστους είναι εθνική αρμοδιότητα. Τα κράτη-μέλη αποφασίζουν πώς ε, θα ε, δομήσουν το δικονομικό σύστημα. Υπάρχει οδηγία για την εναρμόνιση των ε, κανόνων αστικής δικονομίας. Είναι κάτι που δεν είναι εύκολο οφείλουμε να ομολογήσουμε. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάποιο σχέδιο για την ε, εξομάλυνση του κόστους δικαστικών δαπανών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σημαντικό όμως είναι ότι εδώ δεν γίνεται μόνο λόγος για δικαστικές δαπάνες. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Όταν ένας οποιοδήποτε πολίτης ε, θέλει να προσφύγει στο δικαστήριο για την επίλυση ενός θέματος, αυτό συνεπάγεται πολύ υψηλό κόστος. Και, για παράδειγμα, ε, ασφάλιση, έξοδα, έξοδα δικηγόρου. Υπάρχουν πολλές πτυχές, λοιπόν, του συστήματος. Και αυτή τη στιγμή αυτό καθιστά την κατάσταση πολύ δύσκολη. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορούν να γίνουν πάρα πολλά. Ο καλύτερος τρόπος επίλυσης του προβλήματος αυτού είναι σε εθνικό επίπεδο. Ορισμένα κράτη-μέλη ενδεχομένως να εμποδίζουν με την νομοθεσία τους τους πολίτες να προσφεύγουν στα δικαστήρια. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε εμείς εδώ. Υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται και ένας από αυτούς πρέπει να αφορά και τα δικαστικά έξοδα. Αλλά η προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρύθμισης του θέματος αυτού δεν είναι στις ε, προτεραιότητες της Επιτροπής και θεωρούμε αρμοδιότητα της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους τη Σολεδάδη και στη συνέχεια θα πάρει το λόγο ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καταρχήν ευχαριστώ τους αναφέροντες που έθεσαν το θέμα αυτό επιτάπητος. Λοιπόν, η αποτροπή του να ασκήσει κάποιος ένα θεμελιώδη δικαίωμά του είναι το πρώτο ζήτημα εδώ. Βεβαίως και μπορεί να υπάρχει κάποια δαπάνη δικαστική, κάποιο τέλος. Το θέμα είναι εάν αυτό οδηγεί στο να αποτρέπουμε κάποιον από το να ασκήσει το δικαίωμά του. Το δικαίωμά της πρόφασης στη δικαιοσύνη. Και βεβαίως υπάρχει το θέμα της αναλογικότητας. Διότι το θέμα του κατά πόσο είναι λογικό ή όχι δημιουργεί αυτή την αμφισημία του κατά πόσο είναι δύσκολη πρόσβαση στα διάφορα κράτη-μέλη. Βεβαίω και πρέπει να μείνει ανοιχτή η αναφορά, είναι σημαντική, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί. Ξέρω ότι η Κομισιόν το κάνει αυτό, αλλά χρειαζόμαστε και μία έκθεση από την Γιούρη ε, και από την Ένβη, που και αυτή ασχολείται με την προστασία των καταναλωτών, για να δούμε τι πρωτοβουλία θα μπορούσαμε να πάρουμε από εκεί και πέρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ σημαντική την αναφορά, διότι θίγει ένα σοβαρό ζήτημα, όπως είναι το θέμα της δίκαιης δίκης και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Ε, μου κάνει εντύπωση για αυτά που λέει η Κομισιόν, διότι ξεχνάει τελείως τον ε, ε, χάρτη θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το θέμα της δίκαιης δίκης και της πρόσβασης της δικαιοσύνης, στη δικαιοσύνη είναι σημαντικά και υποτίθεται ότι πρέπει να προστατεύονται. Όταν λοιπόν ε, έχουμε σε ένα κράτος μέλος την επιβολή υψηλών δικαστικών εξόδων, τελών και άλλων έτσι, χρηματικών καταβολών με αποτέλεσμα στην πράξη να μην μπορεί κανείς να προσφύγει στη δικαιοσύνη, τότε προκύπτουν θέματα παραβίασης και του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, αν έχουμε και νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτών, όπως έχουμε προκειμένο, που σαφέστατα έχει άμεση σχέση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε εδώ με τον τρόπο της επιβολής υψηλών τελών στην πράξη απαγορεύεται κανείς να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Εγώ θεωρώ λοιπόν σημαντικό αυτό και πιστεύω ότι η Κομισιόν πρέπει να το δει το θέμα αυτό. Όχι μόνο για την Ισπανία. Θα σα φέρω ένα παράδειγμα για την Ελλάδα. Στην Ελλάδα η, τα δικαστικά τέλη διαμορφώνονται με τον νόμο 4446 του 2016. Εν ώψη του ότι μειώνονται συνεχώς οι μισθοί και οι συντάξεις, τα ποσά τα οποία πρέπει να καταβάλει ένας συνταξιούχος για να προσφύγει κατά της μείωσης των συντάξεων, που γίνεται ακόμη και τώρα με τον νέο νόμο που θα έρθει στην εφαρμογή του τετάρτου μνημονίου, μειώνονται ξανά οι μισθοί και οι συντάξει. Τα ποσά τα οποία του ζητούνται είναι δυσανάλογα σε σχέση πλέον με τι συντάξει που παίρνουν. Άρα λοιπόν είναι ένα σοβαρό θέμα παραβίαση τη Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στην Ελλάδα. Δεύτερο θέμα, ακόμη πιο σημαντικό. Α, στα θέματα περί δίκης γύρω από τι φορολογίε. Εάν σου έχει επιβληθεί μια φορολογία α πούμε 20.000 ευρώ, και αμφισβητείς ότι πρέπει να το πληρώσεις, τότε για να κάνεις προσφυγή πρέπει να προκαταβάλεις το 50% της φορολογικής οφειλής, δηλαδή 10.000 ευρώ, συν τα δικαστικά έξοδα. Καταλαβαίνετε ότι στην πράξη κανείς πλέον δεν μπορεί να προσφύγει κατά αποφάσεων των φορολογικών αρχών οι οποίες σου επιβάλλουν ένα ποσό φορολογίας εισοδήματος. Μάλιστα αν σου επιβάλλουν και πρόστιμα και τέλη τότε είναι αδύνατο να προσφύγεις. Άρα λοιπόν απευθύνομαι στην Κομισιόν και φαντάζομαι ότι ακούει αυτά τα οποία λέμε. Το θέμα για μένα είναι σοβαρό. Φυσικά πρέπει να μείνει ανοιχτή η αναφορά. Φυσικά συμφωνώ με την συνάδελφο την Καπεθόν ότι πρέπει να στείλουμε το θέμα στη ΛΥΜΠΕ, διότι είναι ένα θέμα σοβαρό και στη Γιούρη ενδεχόμενα. Αλλά θα ήθελα την Κομισιό να ξαναδεί το ζήτημα τη αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδίω ω παραβίαση τη αρχή τη αναλογικότητα και φυσικά του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων σε σχέση με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και τη δίκαιη δίκη. Επομένως, ε, νομίζω ότι πρέπει να μείνει ανοιχτή και να δούμε παρακάτω πώς θα συνεχίσουμε σε αυτή την υπόθεση. Φαντάζομαι θα έχετε και άλλες υποθέσεις τέτοιες, κυρία Πρόεδρε, και θα έρθουν εδώ, εν ώψη του ότι πλέον αδυνατούν οι πολίτες ε, λόγω υψηλών δικαστικών εξόδων και στην Ελλάδα, ιδίως δεν στην Ελλάδα, να προσφύγουν πλέον κατά των αυθαίρετων αποφάσεων της κυβέρνησης και της Τρόικας που μειώνουν μισθούς συντάξεις και επιβάλλουν πλέον μια φορομπηχτική πολιτική και μια φορολαϊλασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Στανόκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αναφέροντες. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα αυτό. Όχι μόνο για την Ισπανία, αλλά όπως βλέπω και για πολλά άλλα κράτη-μέλη Αναρωτιέμαι γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται τόσο πολύ χρόνο για να κάνει αυτή τη μελέτη. Έπρεπε να εξετάσετε μόνο τη συγκεκριμένη νομοθεσία των κρατών μελών. Η αναφορά είναι αρκετά παλιά και ο κανονισμός ο ίδιος είναι από το 2015 και 2017 αντίστοιχα. Βέβαια, καλωσορίζουμε την απάντησή σας και θα ήθελα μία παράκληση να κάνω να επιταχύνετε ε, τη δουλειά. Και φυσικά θα ζητήσω και εγώ να παραμείνει ανοιχτή αναφορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βαλίνα. Ευχαριστώ Σεσίλη. Εγώ δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τους συναδέλφους που πήραν το λόγο προηγουμένως. Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι ένα δικαίωμα, δεν είναι κάποιο προνόμιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον αναφέροντα, διότι ιδιαίτερα στη χώρα μας ενώ έχουμε πολιτικές λιτότητας, περικοπών, αύξηση της ανεργίας, ε, πάνω από 50% ανεργία των νέων, πολύ εντυπωσιακά στοιχεία, έχουμε δικαστικές δαπάνες ε, οι οποίες όπως πολύ σωστά εξηγήθηκε ξεπερνούν το 50% του ελάχιστου μισθού στη χώρα μου. Ούτε ένας εργαζόμενος δηλαδή μπορεί να προσφύγει κατά μιας απόλυσης παραδείγματος χάρη. Είναι, πρόκειται για μια πραγματική διάκριση και πρέπει να το πούμε σαφώς. Έγινε μια μεταρρύθμιση η οποία ήταν ταξική, είχε ταξικό χαρακτήρα κάποιοι που έχουν χρήματα μπορούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και κάποιοι που δεν έχουν δεν μπορούν. Είναι λοιπόν πολύ σοβαρό το ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα επί του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επιταχύνει τη διαδικασία, διότι όπω βλέπουμε ε, δεν είναι μόνο στη χώρα μα αυτό, αφορά και άλλε χώρε. Και είναι θεμελιώδε δικαίωμα. Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι δικαίωμα που έχουμε όλοι, όχι προνόμιο. Η δικαιοσύνη είναι δωρεάν και είναι καθολική για όλους. Ευχαριστώ. Ρώσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους ε, αναφέροντες. Το είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν υπάρχει εναρμόνιση σε ό,τι αφορά ε, τις δικαστικές δαπάνες. Ούτε προβλέπει η Κομισιόν κάτι τέτοιο. Βεβαίω, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην ομολογία του μιλάει για ισοδυναμία μιλάει για αναλογικότητα πιο συγκεκριμένα. Το είπε και η Σολεδά βέβαια, είναι κάπως ασαφής ο όρος αυτός, όμως δεν πρέπει τα τέλη αυτά ε, να καθιστούν αδύνατη την άσκηση του δικαιώματος. Ε, από ό,τι φαίνεται έχει κλείσει η, έκ, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ θα ήθελα να ξέρω τι λέει αυτή η έκθεση ε, σε ό,τι αφορά τα 28 κράτη-μέλη ε, σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε και πώς ερμηνεύει η Κομισιόν. Έχουμε εδώ ε, καταχρηστικές, ε, καταχρηστικά τέλη, καταχρηστικές δαπάνες ή όχι. Εγώ συμμετέχω και στην Επιτροπή Γιούρη, θα μπορούσαμε να το δούμε το θέμα εκεί, αλλά το πρώτο που θέλουμε, ε, που θα μας ζητήσουν εκεί, είναι πληροφορίες. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορούμε να ακολουθήσουμε και εμείς την οδό που αρμόζει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των ομιλητών. Θα δώσω το λόγο ξανά στον αναφέροντα. Ακούσατε τις απόψεις που εξέφρασαν οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ίσως θα θέλατε εσείς να προσθέσετε κάτι. Ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας. Εσείς ως εκπρόσωποι των πολιτών της Ένωσης πρέπει να γνωρίζετε ότι αφορά την προστασία των καταναλωτών. Το πρόβλημα συχνά δεν έχει να κάνει με την νομοθεσία έχει να κάνει με την εφαρμογή της. Τα εμπόδια, τα διαδικαστικά που αντιμετωπίζει ένας καταναλωτής. Ένα από τα μεγάλα ζητήματα προστασία του καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να κάνει με τις διαδικασίες. Τις διαδικασίες που οδηγούν στην εφαρμογή στην πράξη ε, της προστασίας των καταναλωτών για να μπορέσουμε δηλαδή, να φτάσουμε στην πραγματική προάσπιση των δικαιωμάτων. Οι καταναλωτέ, στο μεγαλύτερο στην τρική ψηφία του, δεν είναι δεθειμένοι να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα δικαστικά προβλήματα. Δεν μπορούν. Χρειάζεται λοιπόν μια μεγαλύτερη εναρμόνιση στι διαδικασίε αυτέ που θα εξασφαλίζουν την προάσπιση των δικαιωμάτων που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για του καταναλωτέ. Πρέπει να υπάρχει μια νέα αναρμονισμένη διαδικασία στο επίπεδο Ένωση που να αφορά αποκλειστικά του καταναλωτέ με μια εναλλακτική διαδικασία σχέση με αυτή που προβλέπεται στην Εθνική Νομοθεσία και θα πρέπει να προωθήσουμε τη χρήση και των ευρωπαϊκών διαδικασιών που υποχρησιμοποιούνται και μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι καταναλωτές τις ε, αιτήσει του ε, όπως ε, μια σειρά από διαδικασίες που στο ευρωπαϊκό επίπεδο που δεν είναι γνωστές πρέπει βέβαια τους άλλους να βελτιωθούν αυτές τις διαδικασίες έτσι ώστε η, η περιπλοκότητα των διαφόρων ε, εντύπων που πρέπει να συμπληρωθούν να μην αποτρέπουν ακόμα περισσότερο τους ε, καταναλωτές. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούν να έχουν πρόσβαση, να μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό και το, να υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που να το επιτρέπει. Να υπάρχει μια εναρμόνιση που να καταργεί αυτές τις δαπάνες στις δικαστικές και του καταναλωτέ όταν προσπαθούν να ασκήσουν τα δικαιώματά του. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω πως είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Συμφωνούμε όλοι πως πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ε, εξήγησε ότι η μελέτη διεξάγεται αυτή τη στιγμή, είναι σχεδόν έτοιμη. Ας μην περιμένουμε λοιπόν ήδη να ολοκληρωθεί η δουλειά της Επιτροπής. Νομίζω πως ε, αφήνουμε λοιπόν ανοιχτή την αναφορά και θα περιμένουμε την παρουσίαση της μελέτης. Και πρέπει να διασφαλίσουμε άρση των εμποδίων αυτών. Δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια για τους πολίτες που θέλουν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα στείλουμε την αναφορά στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για να αποφασίσουν αν θα κάνουν κάτι παραπάνω. Θα θέλετε το λόγο. Ναι, ναι, αν μου επιτρέπετε υπάρχουν κάποια να ερωτήματα και θεωρώ πως ε, πρέπει να τα απαντήσω. Καταρχάς, η μελέτη δεν αφορά μόνο τα δικαστικά έξοδα, αφορά την ε, προστασία και το δικονομικό δίκαιο, προστασία των καταναλωτών στην Ένωση. Βλέπετε εδώ ότι αυτό μόνο που κρατάω αφορά τα δικαστικά έξοδα. Το Ινστιτούτο Max Planck στο Λουξεμβούργο έχει αναλάβει τη μελέτη. Συμμετέχουν έγκριτοι επιστήμονες από όλη την Ευρώπη. Δεν λοιπόν ασχολούμαστε μόνο με τα δικαστικά έξοδα, αλλά γενικότερα. Ε, ε, τον διάμεσο πόρισμα είναι, ε, αυτό λοιπόν δεν συμμερίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά ανάγκη τα αποτελέσματα της μελέτης, αλλά να πω πως Είχα, είχε τον Ινστιτούτο Max Πλάνκα ένα χρόνο για να διεξάγει αυτή την έρευνα, για να κάνει τη μελέτη στα 28 κράτη-μέλη. Τα αποτελέσματα λοιπόν θα τα μάθετε σύντομα. Και κάτι άλλο, να διευκρινίσω ότι δεν υπάρχει καμία διαφωνία ε, στο ότι πρέπει να δράσουμε, πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες που θέλουν να ασκήσουν τα, τα δικαιώματά τους και να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Καταρχάς υπάρχουν νομικά εμπόδια που πρέπει να έρθουν Και μετά τα πρακτικά εμπόδια. Όπως ε, θα δείτε και στην απάντησή μας, Με συγχωρείτε μέχρι να το βρω. There has, okay. There has been έχουν γίνει προσπάθειες εναρμόνισης των δικαστικών εξόδων, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να γίνει αυτό και να συμφωνήσουν όλα τα κράτη-μέλη. Στην πράξη, λοιπόν, δεν θα είναι εύκολο κάτι τέτοιο. Αλλά πόσο μπορούμε στην πράξη να βρούμε ένα σύστημα που θα συμπεριλαμβάνει τα συστήματα όλων των κρατών μελών. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. ο πιο αποτρεπτικός παράγοντας για έναν πολίτη να ασκήσει τα δικαιώματά του να προσφύγει στο δικαστήριο δεν είναι τα δικαστικά έξοδα, είναι τα έξοδα του δικηγόρου. Αυτό βέβαια δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τέλος, ε, όλα τα κράτη-μέλη ζήτησαν ε, στατιστικά στοιχεία από τα Υπουργεία Δικαιοσύνης, αλλά η αλήθεια είναι πως δεν ξέρουμε ακόμα, δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Θα θέλαμε να μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, αλλά δυστυχώς ε, δεν έχουμε. Γι' αυτό λοιπόν ε, στο χέρι των κρατών μελών είναι να μας στείλουν αυτά τα στοιχεία για να μας βοηθήσουν. Σας ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινήσεις. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στη δουλειά, στο έργο σας. Για τα, την ανάλυση των δικονομικών εμποδίων και για θέματα πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Μάλιστα λοιπόν, σας περιμένουμε και για να συνεχίσουμε τον ε, διάλογο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ ε, που ήρθατε εδώ. Ελπίζουμε να βοηθήσαμε και σίγουρα θα είμαστε σε επαφή μέσω της γραμματείας με εσάς. Καλό ε, ταξίδι, καλή επιστροφή στη χώρα σας. Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο. Ο κύριος Μαρια ζήτησε να αναβληθεί η αναφορά 0663 για ε, την επόμενη φορά. Η επόμενη αναφορά είναι 0538 για την καταπολέμηση της τοκογλυφίας εκ μέρους τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο αναφέρον δεν είναι παρόν, όμως θα δώσω το λόγο αμέσως στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους. Κατανοώ ότι θα ασχοληθούμε με δύο αναφορές για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε απαντήσεις στο παρελθόν και οι δύο αφορούν το επίπεδο των επιτοκίων. Μία Ιταλική και μία Κυπριακή αναφορά. Η Ιταλική αναφορά ασχολείται με το επίπεδο των επιτοκίων εφόσον μπορεί να θεωρηθεί το επιτόκιο τοκογλυθικό, ενώ η κυπριακή αναφορά αφορά το επίπεδο των επιτοκίων που αυτή τη στιγμή χρεώνονται στους Κυπρίους καταναλωτές όταν προσπαθούν να πάρουν ένα υπόθηκο δάνειο. Εδώ λοιπόν να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ ε, ευαίσθητη στα θέματα των επιτοκίων. Γι' αυτό, λόγου χάρη, συμπεριλάβαμε στην οδηγία για τα ανυπόθηκα δάνεια και τα καταναλωτικά δάνεια ακριβώς κάποιες ε, απαιτήσει για την αποκάλυψη στοιχείων ώστε οι καταναλωτές προτού υπογράψουν τη σύμβαση να ξέρουν τι ακριβώς τους προσφέρεται και τι ακριβώς υπογράφουν. Επίσης ισχύει η οδηγία για τους ε, αδίκους όρους τους συμβατικού όρου που σκοπό έχουν να προστατεύσουν τους καταναλωτές από άδικου ε, όρου που μπορεί να υποκρύπτονται σε μια σύμβαση και αυτό που δεν κάνουμε ακόμα με την νομοθεσία είναι προφανώ να ρυθμίσουμε το επίπεδο των επιτοκίων αυτό καθεαυτό. Κανείς δεν θα περίμενε να κάνουμε κάτι τέτοιο σε μια οικονομία της αγοράς και της κοινωνίας ταυτόχρονα. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα περάσουμε σύντομα στην εξέταση των λεπτομεριών. Υπάρχει το θέμα του ανταγωνισμού, ανταγωνισμού ε, στα επιτόκια μεταξύ των πιστοτικών ιδρυμάτων. Γι' αυτό λόγου χάρη στην οδηγία των ενυπόθηκων δανείων προβλέψαμε το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο για τους μεσολαβητές δανειοδότες. Με το διαβατήριο αυτό ελπίζουμε ότι στο μέλλον περισσότεροι αλλοδαποί ε, διάμεση για τις πιστώσεις θα προσφέρουν πιστώσεις στα κράτη-μέλη και προσφάτως εγκρίναμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα δράσης για τους καταναλωτές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνει και 12 συγκεκριμένες δράσεις με την πρόθεση να αναθεωρηθεί γενικότερα και ό,τι ισχύει για τα καταναλωτικά δάνεια. Τώρα για την Ιταλική υπόθεση περισσότερο, ο κύριος Λάπη από την Ιταλία έχει παραπονεθεί και υποβάλει αναφορά για το νόμο που αναθεωρήθηκε το 2011 στην Ιταλία και ε, αφορά την τοκογλυφία. Θεωρεί ότι εξαιτία αυτού του νόμου τα επιτόκια έκτοτε εφαρμόζουν και σε αυτά ισχύει μια τέτοια ανώτατη οροφή που διπλασιάστηκε ακριβώς εξαιτία του νέου νόμου, της μεταρρύθμισης αυτής. Ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δηλώσει ότι το άρθρο 2 του νόμου 108-96 της Ιταλικής νομοθεσίας είναι αντισυνταγματικό και ότι παραβιάζει τις ε, βασικές διτάξεις των ευρωπαϊκών συνθήκων. Εξηγήσαμε ήδη στην απάντησή μας και ήδη στην Επιτροπή το 2009 και 2010 είχαμε μια μελέτη για τους περιορισμούς ε, των επιτοκίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μια μελέτη που δίνει μια συνολική σφαιρική εικόνα για το τι είδους περιορισμοί στα επιτόκια εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο. Γιατί σε ευρωπαϊκό δεν υπάρχουν ε, περιορισμοί στα επιτόκια. Η εικόνα που σκιαγραφείται είναι ιδιαίτερα ποικιλόμορφη. Οι ορισμοί είναι πολύ διαφορετικοί. Τα επιτόκια και τα επίπεδά τους, αυτά που χρεώνονται, είναι πολύ διαφορετικά. Το ίδιο και απαντήσει που δίνουν τα κάτι μέλη. Η Ιταλία είναι μία από τις χώρες που το όντι έχει προβλέψει ένα τέτοιο ανώτατο όριο. Η μεθοδολογία μας έχει δεχθεί επικρίσεις, ιδίως μετά την αναφορά. Εφόσον πρόκειται για εθνικό νόμο και εθνική μεθοδολογία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε θέση να το σχολιάσει. Όπως ε, προείπα, το ανώτατο όριο είναι απλώς ένα γενικό πλαίσιο. Δεν φαντάζομαι ότι όλοι οι νόμοι στην Ιταλία ε, φτάνουν ή τέλος πάντων είναι τόσο κοντά στο ανώτατο όριο. Η μόνη συνταγή που βλέπω εδώ είναι περισσότερος ανταγωνισμός, περισσότεροι φορείς και δρόντες σε αυτό το πεδίο Και πολύ γρήγορα να έρθω στην αναφορά του Κυπρίου πολίτη. Δεν το βλέπω σκόπιμο, διότι έχουμε εδώ τον αναφέροντα. Και βάσει των κανόνων θα παρουσιάσει ο ίδιος την υπόθεσή του, μόνος του. Μετά μπορείτε να το απαντήσετε. Ολοκληρώσατε για την πρώτη αναφορά την Ιταλική περίπτωση. Πολύ ωραία. Τώρα λοιπόν θα δώσω τον λόγο για την αναφορά αυτή μιας και αναφέρον λύπη. Να ξεκινήσει η συζήτηση, εφόσον έχει κάποιος κάτι να πει. Κυρία Εύη, ζητήσατε τον λόγο και εσείς, μάλιστα. Πρώτα απ' όλα, πρώτα απ' όλα η κυρία Εύη. Ευχαριστώ που παίρνω το λόγο πριν από τον συνάδελφο. Τον... Ε, μάλλον μπορώ ευχαρίστω να δώσω το λόγο στον συνάδελφο, τον Μάρκο Βάλλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το θέμα αυτό πραγματικά ε, είναι κάτι που με αφορά ιδιαίτερα γιατί είμαι και μέλο τη Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων για την τοκοκληφία. Όντω, έχουμε πρόβλημα στην Ιταλία διότι εφαρμόζεται από το 2011 αυτό ο νόμο. Ο νόμο ο οποίος έχει αυξήσει το όριο που θεωρείται το κογλυφικό. Ακριβώ επειδή υπήρχε ιδιαίτερη πίεση στι αγορέ και οι τράπεζε είχαν μεγάλε δυσκολίε για να αντλήσουν χρήματα και να τροφοδοτήσουν την αγορά. Είχαν ανάγκη λοιπόν από ένα νόμο που να τι εξυπηρετεί. Η τεχνική εξήγηση ήταν αυτή που λάβαμε και από πολλού ε, εμπειρογνώμονε κιόλα προωτήσαμε. Αυτή τη στιγμή Ε, βλέπουμε ότι το φαινόμενο που προκλήθηκε κάπως έχει συγκατηθεί. Όμως είναι εγκληματικό αυτός ο νόμος, γιατί συνεχίζει να εφαρμόζεται. το όριο της οικογλυφίας αυξήθηκε και όταν μιλάμε για επιτόκια τόσο μεγάλα όπως αυτά που επιβάλλουν οι τράπεζες και μπορούν να διατηρούν σε πολύ ψηλά επίπεδα τα επιτόκια, ε, γιατί το όριο από πάνω από το οποίο θα θεωρηθεί το κογλυφικό είναι πολύ αυξημένο, είναι μια πολύ ιδιαίτερη πραγματικότητα αυτή που διαμορφώνεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν τη γνωρίζει την πραγματικότητα και σε πολλά θέματα παρεμβαίνει και σε δημοσιονομικά και σε φορολογικά και κάνει συστάσει. Και α μην τι ε, αποδέχονται οι διάφορε χώρε, όμω καλό είναι να ακούγονται αυτά. Ζητώ λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακριβώ ε, βάσει τη ιδιότητά τη να κάνει μια αξιολόγηση του ποια είναι η κατάσταση των επιτοκίων και τι θα έπρεπε να θεωρείται τοκογλυφία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να δώσει συγκεκριμένε κατευθύνσει, κατευθυντήρε γραμμέ σε κάποιε χώρε όπου τα τραπεζικά του συστήματα, όπου τώρα με, την, ε, με το σύστημα ενιαία εποπτεία από την Κεντρική Τράπεζα για τι εθνικέ, ε, εκεί μπορεί να διατυπωθούν κάποιε συστάσει ώστε να αποφύγουμε κάποιε χώρε να εκμεταλλεύονται την κατάσταση για κάποια τραπεζικά συστήματα, να την εκμεταλλεύονται επίση με νόμου που σε κάποιε περιπτώσει θεωρούνται μεν αλλά εφαρμόζονται ε, όπως έγινε στην Ιταλία από το 2011. Σήμερα είναι πολύ κρίσιμες οι συνθήκες. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή θα μπορούσε από αυτή τη σκοπιά να αναλύσει όχι μόνο την κατάσταση στην Ιταλία αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να ε, δώσει ιδέες, προτάσεις, όχι να επιβάλλει τίποτα, αλλά τουλάχιστον να παροτρύνει προς μια εναρμόνιση, για να υπάρξει έστω μια δυνατότητα να ορίσουμε ένα τοκογλυφικό επιτόκιο, πάνω από το οποίο πρόκειται πια για πραγματική χροκέρδια, για κερδοσκοπία ε, εις βάρος των πολιτών μέσω των δανείων που μπορεί να έχουν ε, πάρει. Εδώ λοιπόν ε, είναι λογικό οι πολίτε να παραπονούνται εδώ ε, παρά την Ευρωπαϊκή Ένωση υποβάλλοντα αυτέ τι δίκαιε αναφορέ. Ευχαριστώ, αλλά έκανα εγώ λάθο εδώ πέρα γιατί δεν σα αναγνώρισα. Δεν κατάλαβα ότι είσαστε μέλο τη Επιτροπή. Τα μέλη τη Επιτροπή έχουν το λόγο πρώτη. Η Ελεονόρα σα παραχώρησε τη θέση τη. Ε, παραχώρησε τη θέση τη υπέρ ημών. Έχετε δίκιο λοιπόν. Ο κύριο Κύριο. Τσίριο. Κύριε Τσίριο. Έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Ναι, είναι ένα θέμα σοβαρό και ιδιαίτερα ευαίσθητο. Και αφορά και τον ιδιωτικό βίο των πολιτών. Οι σχέσεις με τις τράπεζες δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά αφορά τους εργαζομένους και τις οικογένειές, του. οικογένειές τους. Είναι ένα θέμα λοιπόν πολύ ευρύ. Εδώ, στην απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μου φαίνεται ότι υπάρχει μια σοβαρότατη ένδειξη διότι πρέπει να δούμε και το περιεχόμενο των αναφορών μεν, αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε και για την αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το θέμα που κάθε φορά μα απασχολεί. Είναι λοιπόν προφανέ ότι εδώ πρόκειται για ένα σοβαρό και ευαίσθητο θέμα. Από την άλλη, είναι επίση ε, προφανέ ότι πρόκειται για ένα θέμα που είναι αυστηρό τη αρμοδιότητα των ίδιων των κρατών μελών. Εύχομαι λοιπόν να παραμείνει και εθνική αρμοδιότητα σε κάθε περίπτωση. Και είναι λίγο περίεργο εδώ που κάποιε φορέ ε, παραπονιόμαστε για την παρεμβατική Ευρώπη μεν και από την άλλη εδώ σε αυτή την Επιτροπή ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάει στα κάτι μέλη και να του κάνει συστάσει, να του πει να εφαρμόσουν. Το αντίθετο από αυτό που μου φαίνεται ότι συχνά για όμως το θέλουμε να κάνουμε. Μια Ευρώπη που να παρεμβαίνει λιγότερο στη ζωή και την ανεξαρτησία των επιμέρου κατ' μελών. Θεωρώ λοιπόν ότι επειδή πρόκειται για ένα θέμα εθνική αρμοδιότητα, όσα υπόθηκαν είναι πολύ σημαντικά. Η απάντηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θεωρώ ότι ήταν ε, πλήρη και διεξοδική και από τη δική μα την πλευρά η αναφορά αυτή μπορεί να θεωρηθεί ε, ότι έχει εξεταστεί, να λήξει. Βεβαίω, μετά από όσα είπε και ο συνάδελφο που προηγήθηκε, θα μπορούσαμε να δείξουμε επικοδομητικό πνεύμα και να υπάρξει ίσω μια σύγκριση των επιτοκίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάτι που θα μπορούσαμε να το δούμε και με αφορμή την, ερχόμενη, την επόμενη αναφορά. Για λόγου και οικονομία των εργασιών αυτή τη Επιτροπή. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ξανεποβάλουμε αυτό που είπε ο συνάδελφο για την επόμενη αναφορά. Και να καλυφθεί και το θέμα των δικών μα των αρμοδιότητων. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε την εξέταση τη αναφορά αυτή. Η κυρία Εύη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Παρεμβαίνω και εγώ με αφορμή την αναφορά αυτή και το θεωρώ σημαντικό να πάρω τον λόγο γιατί και εμένα μου κάνει κάτι να ακούω ένα από τα μέλη του ΕΛΚ, της Ευρωπαϊκής Ομάδας που είναι πιο φιλευρωπαϊκή αυτού του κοινοβουλίου, να μας λέει για μεγαλύτερη ανεξαρτησία από πλευρά των κατομελών. Αυτό που για μένα σημαίνει ότι καταλήγει η συζήτηση να είναι πάλι το αν θέλουμε λιγότερη ή περισσότερη Ευρώπη. Το καταγγέλουμε εδώ και καιρό αυτό στην Ιταλία το σύστημα των ε, πιστώσεων και των δανείων έχει ε, ευνοηθεί πάρα πολύ από το σύστημα των κανόνων που διαρκώς εξυπηρετεί τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιτρέποντας αυτό που ακριβώς έφτασε να μας καταγγέλει σήμερα ο αναφέρον, με επιτόκια τα οποία είναι σε ψηλότατα επίπεδα. Να θυμίσω εδώ και τις πολυάριθμες αυτοκτονίες που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια μεταξύ των οποίων ε, περιλαμβάνονται πολλοί επιχειρηματίες οι οποίοι καταστράφηκαν από, τις, ε, από τα επιτόκια που επιβάλλουν οι τράπεζες. Σε πλήρη ασυδοσία με πλήρη ε, αποτυχία των εποπτικών φορέων που δεν κατάφεραν να ελέγξουν τίποτα στην Ιταλία. Τα, ε, τους φορείς αυτούς του ελέγχου και της εποπτείας τους κατέχουν ιδιώτες. Οπότε επαναλαμβάνεται ο μηχανισμός του ελέγχου που επανελέγχει τους ίδιους και τους ίδιους. Οι πολυάριθμοι πολίτες που οργανώθηκαν σε κινήματα και ενώσεις πολλές φορές ευαίσθησαν στην προσοχή των δικαστών τη δράση των τραπεζών χωρίς να παραδεθούν τα όπλα. Και πολλέ φορές μάλιστα οι τράπεζε θεωρήθηκαν ένοχε για την τοκογραφική του δράση και αναγκάστηκαν να υποβάλουν ε, αποζημιώσει στους πολίτες. Εμείς ως κίνημα πέντε αστέρων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στο εθνικό ζητούμε μια ριζική μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού και τραπεζικού μας συστήματος να υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των δραστηριοτήτων ε, ε, κλασικής δανειοδότησης και των κερδοσκοπικών δράσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακούσαμε, δεν έχει και πολλά, θέματα, πολλά στοιχεία να παρατηρήσει επί της ουσίας. Διότι εκεί που έχει αναλάβει δράση έχει προκαλέσει ανυπολόγιστε καταστροφέ. Ελπίζω οι ριζικέ μεταρρυθμίσει που θα γίνουν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο να γίνουν στο δυνατόν συντομότερα. Και εγώ ζητώ η αναφορά αυτή να παραμείνει ανοιχτή, γιατί το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο και πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη να το ξαναδούμε και στο μέλλον. Για να αποτιμήσουμε πώ θα έχει διαμορφωθεί τότε η κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Για το μέλλον, λοιπόν, και για το υπόλοιπο σημερινό απόγευμα. Ε, παρακαλώ, εάν υπάρξουν Ιταλοί συνάδελφοι που θέλουν μια προσωπική βεντέτα μεταξύ τους, να φύγουν από την αίθουσα και να λύσουν τα θέματα εκτός. Θα ήταν πολύ καλό αυτό για όλους μας και θα ε, ήθελα να αποφύγουμε να γίνονται δηλώσει κατά των άλλων πολιτικών ομάδων που βρίσκονται στην αίθουσα, γιατί ε, κυκλοφορούμε και ακουγόμαστε και στο διαδίκτυο. Δεν είναι πολύ ωραίο να λύνετε τα εσωτερικά σα ζητήματα εδώ. Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, δεν έκανα καμία δήλωση ε, απευθεία κατά άλλη πολιτική ομάδα ή κόμματο. Ήταν μια γενική δήλωση ω ε, πολιτικού κόμματο που είμαστε εδώ στο Κοινοβούλιο ακριβώ για αυτόν τον σκοπό. Ήταν ευρωπαϊκού χαρακτήρα η δήλωσή μου. Ναι, είπατε αυτά που είπατε και καταγράφησαν. Α προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε την εξέταση αυτή τη αναφορά. Η μόνη πρόταση ήταν να παραμείνει ανοιχτή. Το επιθυμεί αυτό και η υπόλοιπη επιτροπή. Α, εσείς δεν το είπατε αυτό. Εγώ θα ήθελα να κλείσει να δούμε τι θα κάνουμε με αυτήν την αναφορά. Να στείλουμε μια επιστολή λοιπόν στον αναφέροντα, όπου θα συμβουλεύουμε να υποβάλει την αναφορά του είτε στην Τράπεζα της Ιταλίας ή στον ε, υπεύθυνο διαμεσολαβητή για τα χρηματοπροστατικά και τα οικονομικά που μόλις διορίστηκε και θα το πούμε πώς να το κάνει αυτό με τα σχετικά link της ε, ανάλογης διευθύνσης στο ίντερνετ και να κλείσουμε την αναφορά. Αυτό θα επιθυμούσα να κάνουμε. Να το κάνω φαίνεται ότι ναι, υπάρχει διαφορετική άποψη από τους πέντε αστέρες από ό,τι φαίνεται, αλλά νομίζω ότι κατά τα άλλα υπάρχει πλειοψηφία. Να προχωρήσουμε όπως είπα. Ας το κάνουμε λοιπόν αυτό και ας περάσουμε στην επόμενη αναφορά, η οποία είναι είναι 17-21, ενό συναδέλφου, το κύριο Τάκη Χατζηγεωργίου από την Κύπρο. Αφορά τα εξαιρετικά υψηλά επιτόκια που χρώνουν οι τράπεζε στην Κύπρο. Τώρα, ακούστε με προσεκτικά διότι ο συνάδελφος παρίσταται. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ. Ήθελα απλώς να θυμίσω σε όλους ότι οι ίδιοι κανόνες που αφορούν ε, τους βουλευτέ ω αναφέροντε είναι αυτοί που σχεδόν για κάθε άλλον άνθρωπο. Ε, δηλαδή η εξή. Ο καθή έχει δικαίωμα σε αναφορά και όταν ο αναφέρον παρουσιάζει το θέμα του στην Επιτροπή, μπορεί να το παρουσιάσει εφόσον είναι ευρωβουλευτή όπω κάθε άλλο αναφέρον. Αυτό εξυπακούεται. Δεν μπορεί όμω να συμμετάσχει στη διαδικασία λήψη απόφαση. Δηλαδή, συζήτηση περί τη αναφορά και κάποιε φορέ και ψηφοφορία για την ίδια την αναφορά. Παρ' όλα αυτά, είστε απολύτω ευπρόσδεκτο να λάβετε το λόγο και να εκφράσετε τι απόψει σα για να αποσαφηνίσετε την δική σα οπτική γωνία περί τη αναφορά σα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν είναι τιμή για κάθε πολιτικό να παρουσιάζει ένα θέμα ως πολίτης. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να αισθάνεται ένας πολιτικός ότι τον αναβαθμίζει. Περαιτέρω, η ισότητα στην αντίκριση πολιτικών ή πολιτών είναι ε, βασικό συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας και της λειτουργίας της ε, Επιτροπής μας. Καταρχήν θέλω να πω ότι ε, έχω εν καλυφθεί σε ζητήματα τα οποία ήθελα να πω και από τον κύριο Βάλη και από την κυρία Εύη. Ένα μεγάλο κομμάτι των επιχειρημάτων μου ε, βρίσκονται στα όσα έχουν ήδη λεχθεί, γι' αυτό ε, θα παραμείνω στα επιπρόσθετα που θα ήθελα να πω. Τα επιτόκια στην Κύπρο, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι και αλλού, θα σταθώ όμως στα της Κύπρου, είναι ληστρικά. Ε, υπερβαίνουν κάθε όριο λογικής. Και η απάντηση της Επιτροπής μάλλον περισσότερες ανησυχίες μου δημιουργεί παρά να μου δείχνει ότι υπάρχει ένας δρόμος επίλυσης των προβλημάτων. Διαβάζω από ένα κομμάτι της απάντησης της Επιτροπής, το οποίο αν είναι καλά τα ελληνικά μου, ε, και είναι, ή αν είναι σωστή η μετάφραση και πρέπει να είναι, ε, μου προσθέτει ε, περισσότερες ανησυχίες. Λέει ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 93 κάθετος 13 το ύψος του επιτοκίου μπορεί να θεωρηθεί ως αμοιβή και κατά συνέπεια το ανάλογο ή μη των υπηρεσιών ή των αγαθών που θα παρασχεθούν ως αντάλλαγμα μπορεί να εξαιρείται από την δικαστική αξιολόγηση κατανοώ σωστά λοιπόν, εδώ λέει ότι όποιο επιτόκιο θέλει μπορεί να βάλει η τράπεζα και δεν μπορεί να πάει ούτε δικαστήριο. Αυτό νομίζω ότι δεν, δεν ε, αγγίζει από οποιαδήποτε σκοπιά και αν το δει κανεί ε, τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών να μπορούν να απευθύνονται σε ανώτερες αρχές ε, και να ζητήσουν το δίκαιο τους. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι και δεν ξέρω αν συμβαίνει σε άλλα κράτη. Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω. Εάν ένας Κύπριος υπογράψει ως εγγυητής για ένα ποσό 50.000 ευρώ για κάποιον άλλο συμπολίτη του, δικαιούται η τράπεζα στην συνέχεια να αυξήσει το ποσό που δανείστηκε ο Β από 50.000 στις 200 και να βρεθείς να είσαι εγγυητής σε ποσό των 200.000 ενώ εσύ υπογράψεις για 50. Αυτό και αν είναι παραβίαση ε, κάθε, κάθε ανθρώπινου δικαιώματος. Ούτε καν ενημέρωση δηλαδή. Μπορεί να το μάθεις ε, πάρα πολύ τυχαία. Λέει επίσης η Επιτροπή ότι με την εφαρμογή της ε, οδηγίας 2014-17 εγκρίθηκε πρέπει να πω εδώ από την Κυπριακή Βουλή μόλις προχτές 24, 28 Τετάρτου εν άρα χρειάζεται επικαιροποίηση η απάντηση της Επιτροπής δεδομένου ότι τώρα έχουμε ε, έγκριση αυτής της ε, ε, οδηγίας. Λέει λοιπόν ότι θα λυθεί το πρόβλημα διότι οι Κύπροι μετά από την εφαρμογή αυτής της οδηγίας αυξάνεται ο ανταγωνισμός και θα δικαιούνται να δανείζονται και από άλλα κράτη. Με συγχωρείτε αλλά <clears throat> εγώ προσωπικά αποτάθηκα σε βελγική τράπεζα εδώ για να δανειστώ και βεβαίω πρέπει να βάλει κάτι ω υποθήκη. Και σου λέει πρέπει να έχει εδώ κάτι στο Βέλγιο. Δεν δέχεται εγγύηση περιουσία που έχει σε άλλο κράτο μέλο. Ποια λοιπόν είναι αυτή η προσπάθεια ενοποίηση των περισσότερη Ευρώπη, όπω λέει το ΕΛΚ, και υπερασπίζομαι εδώ την κυρία Εύη, που είπε πολύ καθαρά ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα <clears throat> ουσιαστικά μα φωνάζει μέρα νύχτα για περισσότερη Ευρώπη, και ξαφνικά εδώ μα λέει εξουσίες των κρατών μελών. Πώς είναι δυνατόν να, να θεωρείτε ότι είναι επιτεύξιμο να κερδίσεις, να πάρεις δάνειο από μια γερμανική τράπεζα όντας Κύπριος από τη στιγμή που θα σου ζητήσει να έχεις περιουσία στη Γερμανία. Νομίζω ότι δεν παρέχει καμιά θεραπεία αυτό το πράγμα. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν βλέπω ότι θα υπάρξει λύση διότι η θεωρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο ανταγωνισμός. Εδώ δεν υπάρχει καν ο ανταγωνισμός τον οποίο προσφέρει ως θεραπεία με την απάντησή της η Επιτροπή, αναφέρομαι στο παράδειγμα που έχω πει πιο πριν, και άρα ουσιαστικά αυτό που λέει είναι ότι οι τράπεζες δικαιούνται, το λέει πάρα πολύ καθαρά, το διάβασα πριν, δικαιούνται να βάζουν οποιοδήποτε ε, επιτόκιο θέλουν και δεν μπορείς να αποταθείς ούτε στο δικαστήριο. Κλείνω ζητώντας να μείνει ανοιχτή η, η αναφορά μου και να ζητήσω από την Επιτροπή να επικαιροποιήσει την απάντησή της δεδομένης της έγκρισης της Οδηγίας 2014 του 17 από το Κυπριακό Κοινοβούλιο στις 28 τετάρτη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα ο λόγος είναι για κύριε Μάρια. Για κύριο Μάρια. Because your, your, your Greek are perfect, but sometimes they need uh, some correction. In any case, I will speak in Greek. Uh, <clears throat> το θέμα το, της αναφοράς αυτής του συναδέλφου Χατζηγεωργίου αλλά και η προηγούμενη αναφορά νομίζω βάζουν τα ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή έχουμε ένα καθεστώς τραπεζοκρατίας όπου πλέον οι τράπεζες επιβάλλουν ιδιαίτερα υψηλά επιτόκια και στην ουσία είναι κράτος εν κράτη. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα. Το δεύτερο συμπέρασμα που έχουμε δει είναι ότι στην τραπεζική κρίση που ήρθε οι πολίτες διέσωσαν τις τράπεζες και αφού οι τράπεζες διασώθηκαν με ανακεφαλαιοποιήσεις και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στα υπόλοιπα κράτη, τώρα επιτίθενται κατά των πολιτών που τις διέσωσαν, διότι οι πολίτες ταυτόχρονα ως δανειολήπτες δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δανειά τους. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο. Το τρίτο θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ο επαρκής, θα έλεγα, έλεγχος από την ίδια την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το τέταρτο σημείο υπάρχει η έννοια της τοκογλυφίας. Η τοκογλυφία είναι προσδιορισμένη και ξεκάθαρη. Και τα δικαστήρια και στην Ελλάδα και σε πολλά κράτη έχουν προσδιορίσει τι είναι τοκογλυφία. Επομένως το να απαντά κανείς ότι το επιτόκιο απλά είναι η ανταμοιβή της τράπεζας για την παροχή των υπηρεσιών δεν προσφέρει επαρκείς απαντήσεις διότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο η τράπεζα να χρεώνει ό,τι θέλει ως επιτόκιο. Αυτό όμως δεν επιτρέπεται διότι οδηγεί στην τοκογλυφία. Το γεγονός ότι δήθεν θα υπάρξει ανταγωνισμός σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι θα μειωθούν τα επιτόκια στην πράξη δεν το έχουμε δει διότι υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια και στο δανειολήπτη να δανειστεί απευθείας από άλλη τράπεζα σε άλλο κράτος μέλος αλλά και από παροχή υπηρεσιών των τραπεζών σε άλλα κράτη-μέλη. Το επόμενο στοιχείο που υπάρχει και το οποίο δεν αναφέρθηκε είναι τα τεράστια προβλήματα όσων έχουν δανειστεί σε ελβετικό φράγκο. Το υπενόησε λίγο η Κομισιόν αναφερόμενη στα δικαιώματα προστασίας του καταναλωτή διότι εκεί δεν έχουμε υπερβολικά επιτόκια, αλλά διαφορά νομίσματος και αξίας του ελβετικού φράγκου σε σχέση με το ευρώ και στην ουσία έχουν φτάσει 70.000 Έλληνες δανειολήπτες, αλλά και σε άλλα μέρη και στην Κύπρο και στη Βρετανία και σε άλλα μέρη να μην μπορούν να πληρώσουν πλέον τα δάνειά τους. Και έρχεται η Κομισιόν πράγματι με μια νομοθεσία να αντιμετωπίσει το θέμα, αλλά για το μέλλον, όχι για το παρελθόν. Και το έχουμε ξαναπεί εδώ ότι κάτι έπρεπε να γίνει αναδρομικά διότι αναδρομικά έπρεπε να λυθεί το πρόβλημα, διότι το έχουν όλοι οι συνάδελφοί μας. Το επόμενο θέμα το οποίο προκύπτει, γιατί εγώ νομίζω ότι είναι σοβαρό το ζήτημα και πρέπει να το δούμε πιο γενικά, με αφορμή τις δύο περιπτώσεις Ιταλίας και της Κύπρου, πρέπει να δούμε γενικότερα, είναι οι ε, ε, τα διάφορα ποσά που επιβάλλουν ως τέλη οι διάφορες τράπεζες. Δηλαδή στην Ελλάδα υπάρχει ένας νόμος ο 128 του 1975 επιβάλλει ένα χαράτσι ουσιαστικά επί του ποσού του επιτοκίου και αυτός ο νόμος υπήρχε για την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών, αυτό τώρα δεν υπάρχει στην πράξη, και όσο καθυστερείς να πληρώσεις, τόσο σου βάζουν συνεχώς αυτό το χαράτσι. Με αποτέλεσμα οι Έλληνες δανειολήπτες που χρωστούν και κάνουν ρύθμιση και πάνε τις δόσεις πιο πίσω, μπαίνει αυτό το επιτόκιο συνεχώς ως ποινή πάνω στη τιμή, στο ποσό που οφείλουν. Γεγονός απαράδεκτο. Και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να το εξετάσουμε. Άρα λοιπόν για να κλείσω κύριε Πρόεδρε. Πρώτον, θεωρώ ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η συγκεκριμένη πλέον αναφορά. Δεύτερον, να υπάρξει μία επιστολή πιστεύω και προς την Κυπριακή κυβέρνηση για να μας πει πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το θέμα. Τρίτον, νομίζω ότι πρέπει να απευθύνουμε μία επιστολή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στον κύριο Ντράγκη, να δει και αυτός τα θέματα που έχουν. Θεωρώ ότι έχει, να μην πω ευθύνε, έχει αρμοδιότητες και υπευθυνότητα η Κεντρική Τράπεζα που πρέπει να δει το ζήτημα τι θα γίνει με την λειτουργία αυτής της κατάστασης. Και επιπλέον και στην οίκον που νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Άρα λοιπόν σφαιρικά μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, να το κρατήσουμε ανοιχτό, να δούμε όλε τι πλευρέ. Είναι σοβαρό το ζήτημα, γιατί υπάρχει επιπλέον και η άλλη πλευρά. Ότι οι τράπεζε πολλούν τα δάνεια στα κοράκια και τα κοράκια, τα, τα επιθετικά funds παίρνουν τα δάνεια σε χαμηλή τιμή με αποτέλεσμα να βγάζουν τα σπίτια στους φυρίς στην Ισπανία, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες στο 1 δέκατον της τιμής. Δηλαδή υψηλά επιτόκια, ο δανειολήπτης δεν μπορεί να πληρώσει και εν συνεχεία τα επιθετικά φαντς αγοράζουν τα δάνεια από τις τράπεζες και τα παίρνουν στο 1 δέκατο της τιμής. Αυτό και αν είναι πλέον εκμετάλλευση. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι σοβαρά τα θέματα και θα πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά. Ευχαριστώ. Και τώρα, για δεύτερη φορά σήμερα, θα στραφώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πω έχετε και πάλι το λόγο, κύριε Στάινερ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εστιάσω εδώ στην αναφορά από την Κύπρο και αυτά που είπε ο κύριος Ευρωβουλευτής από την Κύπρο και ο Ευρωβουλευτής από την Ελλάδα. Στην προηγούμενη τοποθέτησή μου τόνισα την σημασία του ανταγωνισμού. Συμφωνώ απόλυτα με εσάς. Ο ανταγωνισμός καθ' αυτός δεν είναι πανάκια. Χρειάζεται να δούμε τους λόγους για τους οποίους δυστυχώς τα επιτόκια αυτή τη στιγμή στην Κύπρο και ίσως στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα υψηλά παρά τα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια που έχει ως πολιτική Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εδώ σίγουρα υπάρχει περιθώριο κέρδους από τις τράπεζες, αλλά κοιτάξαμε την περίπτωση της Κύπρου. Και από χθες, αν δούμε το ε, spread που χρεώνουν για ένα στεγαστικό δάνειο, ε, ε, το σταθερό επιτόκιο για ένα στεγαστικό δάνειο 5 ετών είναι 6%. Ο καταναλωτής δηλαδή, αυτός που δανείζεται, θα πρέπει να πληρώσει περίπου 6,25% ως επιτόκιο. Αυτό από την Κεντρική Τράπεζα. Και σίγουρα σε σχέση με έναν πολίτη που δανείζεται στη Γερμανία, το επιτόκιο αυτό είναι πολύ ψηλό. Να πω όμως ότι δυστυχώς η Κύπρος μέχρι σήμερα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων. Περίπου 50% των δανείων δεν εξυπηρετούνται. Και στα άλλα κράτη-μέλη το ποσοστό αυτό είναι από 5 έως 7%. Εάν λοιπόν οι τράπεζες της Κύπρου μπορούν να προμηθευτούν φτηνό χρήμα για να δανείσουν και αυτό είναι και το σκεπτικό πίσω από την ε, πολιτική επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να δούμε δηλαδή ε, πώς θα βοηθήσουμε τις ε, μικρές επενδύσεις. Όταν δανείζουν χρήματα, πρέπει να δουν ποιες είναι οι πιθανότητες να πάρουν πίσω τα χρήματά τους σε τακτικές δόσεις. Και αυτό αφορά όλους και εκείνους που μπορούν να πληρώσουν τα δάνεια στην ώρα τους. Εκείνοι δυστυχώς καλύπτουν και αυτούς που δεν μπορούν να πληρώσουν το δάνειο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το εξαιρετικά ψηλό επιτόκιο. Ε, να συγκρίνουμε λίγο την κατάσταση και με την Ιρλανδία, η οποία πέρασε μία παρόμοια κατάσταση. Είχε πολύ, ε, πέρασε πολύ δύσκολη κρίση στον τομέα των ακινήτων. Εκεί Ακούστηκαν και εκεί παράπονα καταγγελίε ότι οι τράπεζε χρεώνουν ιδιαίτερα υψηλά επιτόκια. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοιτάξει. Εμείς κοιτάζουμε τις εκθέσεις για κάθε χώρα, αλλά η Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας αποφάσισε να διεξάγει μία έρευνα για την ανταγωνιστικότητα εντός του τραπεζικού τομέα, έτσι ώστε να δουν εάν τα επιτόκια αυτά είναι αναλογικά του κινδύνου που αναλαμβάνει μια τράπεζα όταν δανείζει ή εάν οι τράπεζες κερδίζουν επιπλέον χρήματα και έχουν κάποιο πρόσθετο κέρδος το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί υπερβολικό. Και σε αυτή την περίπτωση θα πω ξανά πως ε, θα μπορούσαμε να δούμε το θέμα εθνικά, να αντιμετωπιστεί το θέμα σε εθνικό επίπεδο. Εάν μου επιτρέπετε όμως θα ήθελα να σας ενημερώσω και για τι γίνεται σχετικά με την ε, οδηγία για τα στεγαστικά δάνεια στην Κύπρο. Πράγματι, η Κυπριακή Βουλή ενέκρινε στις 28 Απριλίου την οδηγία Η αρχική ημερομηνία έγκρισης ήταν έγκριση πέρασε δηλαδή ένας χρόνος, αλλά η Κύπρος δηλαδη ενα είναι η μόνη χώρα που καθυστέρησε στην εφαρμογή της ε, οδηγίας. Υπάρχουν και άλλες τρεις χώρες, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Κροατία, οι οποίες παραπέμφθηκαν μαζί με την Κύπρο στο ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η Κυπριακή Βουλή βέβαια τώρα ε, ενέκρινε τη μεταφορά της οδηγίας στην νομοθεσία της και ελπίζουμε να υπογραφεί σύντομα, να δημοσιευθεί στην ε, επίσημη εφημερίδα, στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, έτσι ώστε να θεωρηθεί πλήρως ε, εγκεκριμένη. Και μετά θα δούμε τι άλλο θα γίνει με το δικαστήριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις διευκρινήσεις που μας δώσατε. Ο κύριος Τσίριο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέμα παρόμοιο, αλλά και διαφορετικό σε σχέση με την προηγούμενη αναφορά. Διότι επί των λεπτομεριών, εκεί βλέπαμε μία από τις πτυχές της τοκογλυφίας, ενώ εδώ και υπό το φως της παρουσίασης του συναδέλφου ακούστηκαν κάποιες παρατηρήσεις που νομίζω έχουν διαφορετική προέλευση και χαρακτήρα. Δεν είναι απλή ε, αξιολόγηση του πώς λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα δηλαδή. Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιες φορές κατηγορείται ότι θέλει να ε, δολοφονήσει την ανεξαρτησία των κρατών μελών. Λογικό είναι λοιπόν αυτά να την προασπίζονται κάποιες φορές. Εδώ το θέμα είναι και τι προσωπικές εγγυήσεις πρέπει να δίνει κανείς σε μια τράπεζα. Ο εγγυητής είναι εγγυητής για το ποσό το οποίο έχει αναλάβει, για το οποίο έχει αναλάβει ευθύνη. Δεν μπορεί μια τράπεζα να αλλάζει αυτό το ποσό όποτε θέλει, δεν έχει πια να κάνει με τα τραπεζικά, εφόσον υπάρχει τέτοια μεταβολή του ποσού. Έχει να κάνει με τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα ατομικά mm. δικαιώματα. Και μια άλλη παρατήρηση πολύ σημαντική, η δυνατότητα να απευθυνθεί κανείς στις τράπεζες σε άλλων χωρών. Υπάρχει δυσκολία εδώ σε σχέση με τις εγγυήσεις που μπορεί να δώσει κανείς στο εσωτερικό των κρατών και αναλόγως αν ζητά κανείς ένα δάνειο ή ένα στεγαστικό δάνειο. Εδώ νομίζω η ουσία των παρατηρήσεων του συναδέλφου ξεπερνά το τραπεζικό την τραπεζική διάσταση. Είναι ευρύτερης, ευρύτερο, γενικότερο χαρακτήρα. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια σωστή αξιολόγηση για να δούμε πώς οι νέοι κανόνες έχουν εφαρμοστεί στους πρώτους μηνές ζωής τους και θα έλεγα ότι και η δική μας ομάδα συμφωνεί να παραμείνει αναφορά ανοιχτή. Άντζελα. E, και εμεί από πλευρά Γκουέ e ζητούμε να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, διότι εξηγήσει που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εντάξει, τελικά εφαρμόζουμε το ένα το άλλο δόγμα, δόγμα το τι μα συμφέρει. Βεβαίω οι τράπεζε χρειάζονται, εντάξει, υπερασπίζεστε την ελεύθερη, το ελεύθερη αγορά κτλ. Αλλά χρειάζεται και ρύθμιση, χρειάζεται και έλεγχο. Η Ευρώπη έδωσε τόσα χρήματα για τη διάσωση των τραπεζών στην ε, Ισπανία, τη χώρα μου, και την χρέο το πληρώνουν οι πολίτε. Επίση, οι απόλυε μια τράπεζα σχετίζονται και με τα επιτόκια τα επενδυτικά και το που επενδύει τα χρήματά της η τράπεζα. Δεν θα πρέπει λοιπόν ε, να χαλαρώσουμε εδώ, διότι έχουμε πάθη από τις τράπεζες. Έχουμε πάθη από τις εξώσεις, από τα τοξικά προϊόντα. Θα πρέπει λοιπόν να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και θα πρέπει να απευθυνθεί στις αρχές της Κύπρου και της Ιταλίας στην προηγούμενη περίπτωση. Ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι αφού είναι τράπεζα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Όταν κάποιος έχει ένα εμπόριο υπάρχει κίνδυνος, υπάρχει και ρίσκο. Η κυρία Κούνεβα είναι η τελευταία ομιλητρία. Παρακαλώ προσπαθήστε να είστε σύντομοι διότι έχουμε ακόμα μία ε, αναφορά να εξετάσουμε πριν από το τέλος της ημέρας. Στις 6.30 δεν θα έχουμε πια διερμηνία, οπότε πρέπει κάπως να επιταχύνουμε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Το πρόβλημα ε, της Κύπρου αναδεικνύει το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει και στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με την τραπεζική αυτερησία. Τα δάνεια με το ελβετικό φράγκο είναι μια πλευρά του προβλήματος. Στην Ελλάδα δεν θα υπήρχε ο περίφημος νόμος Κατσέλη που έβαλε φρένο στις κατασχέσεις χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες τα είχαν βρεθεί στο δρόμο. Σύμφωνα με τους ε, κυρίους Χατζηγεωργίου και Μαριά να μείνει ανοιχτή η αναφορά και να επευθύνομαι επιστολή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επίσης, προτείνω ακρόαση και έκθεση πρωτοβουλία για όλες τις αναφορές από όλες τις χώρες που έχουν έρθει στην Επιτροπή Αναφορών. Γιατί ξέρω ότι παρόμοιες καταστάσεις υπάρχουν και σε άλλες χώρες και να δούμε το ζήτημα πιο συνολικά και να καταλάβουμε ακριβώς τι προβλήματα έχουμε και να δουλέψουμε ταυτόχρονα τα ζητήματα των χωρών στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Thank you very much. Now, I... Σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, αλλά πρώτα θα δώσω το λόγο στον συναδελφό μας για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, η κύρια κουβέντα που έχω να πω είναι ότι η αναφορά πρέπει να μείνει ανοιχτή. Ε, καμία αμφιβολία επί τούτου. Η αναφορά επίσης εκ μέρους της Επιτροπής που οφείλω να πω ότι ήταν ειλικρινής και αυτό είναι χρήσιμο στη δουλειά μας ότι τα επιτόκια στην Κύπρο είναι 6,25 συν τα τέλη κλπ. Η αναφορά εκ μέρους μου ότι είναι ληστρικά επιτόκια είναι μειώνει τη βαρύτητα του προβλήματος το οποίο συζητάμε. Το τρίτο που έχω να πω είναι ότι πρέπει να πάει επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου που να ζητά σκέψεις, ιδέες, διευκρινήσεις για το πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το ζήτημα και προς την, και προς την ε, Κυπριακή Κεντρική Τράπεζα το ίδιο. Και το τελευταίο ζήτημα που έχω να αναδείξω, να επαναφέρω από την προηγούμενη κουβέντα που έκαμα, είναι ότι πρέπει, μέσα στην επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μπει και μια αναφορά για το πώς μπορεί πρακτικά ένας πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας να μπορέσει να πάρει δάνειο από τράπεζα της Γερμανίας δεδομένου ότι μάλλον δεν του επιτρέπουν να πάρει δάνειο εφόσον δεν έχει περιουσία στη χώρα στην οποία η τράπεζα αυτή είναι εγκατεστημένη, από την οποία θα αιτηθεί δηλαδή το δάνειο. Αυτά και ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε. Θα παραμείνει η αναφορά ανοιχτή. Όπως ε, είπαν και όλοι όσοι τοποθετήθηκαν. Θα κρατήσουμε λοιπόν την αναφορά ανοιχτή και προσμένουμε σε έναν καλό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα στείλουμε και μία επιστολή στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και στην Ένωση Τραπεζών Κύπρου, εκφράζοντας την ικανοποίησή μας για την έγκριση της οδηγίας και εκφράζοντας μεγάλες ανησυχίες για το γεγονός ότι το 50% των ε, μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι ένα τεράστιο ποσοστό, ενώ σε άλλα κράτη-μέλη το ποσοστό αυτό είναι 5-7%. Νομίζω μπορούμε να το αναφέρουμε αυτό ως κάτι που μας προκαλεί ιδιαίτερε ανησυχίε και να ζητήσουμε και τη δική τους άποψη για τη συγκεκριμένη αναφορά. Συμφωνείτε? Σίγουρα. Και μια επιστολή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ναι, και σε ό,τι αφορά την πρόταση της κυρίας Κούνεβα δεν μπορούμε να το κάνουμε, διότι όλα αυτά πρέπει να τα αποφασίσουν οι συντονιστές. Μπορείτε λοιπόν να μιλήσετε με τον αρμόδιο συντονιστή σας, με τους υπεύθυνου πολιτικής και να συζητηθεί σε μια συνάντηση των συντονιστών αργότερα. Και επίσης να σταλεί μια επιστολή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ναι, για την δυνατότητα ή όχι που έχει ένας πολίτης της Κύπρου να πάρει δάνειο από άλλη χώρα. Ναι, θα στείλουμε και σε αυτούς επιστολή. Και εάν επιθυμείτε να γίνει κάποια παραπάνω δράση, παρακαλώ να μιλήσετε με τον αρμόδιο συντονιστή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας περάσουμε στο τελευταίο σημείο για σήμερα, την αναφορά 175 κάθετος 2015 για την εξαίρεση της μηχανικής ε, ταυπή από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων. Ο αναφέρον είναι εδώ, ονομάζεται Πέντρο Ντελατόρε. Θα σας δώσω το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους. Θα είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος ε, είναι λίγος ο χρόνος που έχω στη διάθεσή μου βέβαια από το 2008 και μετά η τεχνική μηχανική στον τομέα της πληροφορική έμειναν ε, σε ένα κενό σύμφωνα με την οδηγία 2005-96 ε, βρέθηκαν εκτός πλαισίου δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες βρέθηκαν στο δρόμο βρεθήκαμε εκτό νομικού πλαισίου και σε ό,τι αφορά την άσκηση του επαγγελματό μα και σε ό,τι αφορά την αναγνώριση των προσόντων μα. Έτσι λοιπόν βρέθηκαν, βρεθήκαμε εκτός του πλαισίου. Ναι, σας παρακαλώ να σας πω ότι ε, οι πληροφορίες μου λένε ότι μιλάτε πάρα πάρα πολύ γρήγορα και δεν θα μπορέσω να διαμαρτύρω την το που λέτε. Προσπαθήστε να τα πείτε λίγο πιο αργά. Ναι, είναι λόγω χρόνου. Ναι, καταλαβαίνω ένα χοντικό, αλλά με, το, με την ησυχία σας. Επαναλαμβάνω βρέθηκαν λοιπόν εκτός του νομικού πλαισίου και για την άσκηση του επαγγέλματο και σε ό,τι αφορά τα προσόντα τους και την αναγνώρισή τους. Μιλάμε για το μοναδικό επίσημο ε, δίπλωμα το οποίο δεν ρυθμίζεται στην Ισπανία. Έτσι λοιπόν κυρίες και κύριοι αυτό σημαίνει ότι η Ισπανία δεν αναγνωρίζει τα προσόντα των τεχνικών μηχανικών στον τομέα της πληροφορικής δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο. Αυτό έχει δύο επιπτώσεις. Πρώτον, οι, οι Ισπανοί επαγγελματίε δεν μπορούν να παρέχουν υπηρεσίε στα κράτη-μέλη ε, όπου δεν υπάρχει ρύθμιση. Επίση, δεν μπορούμε να ζητήσουμε την επαγγελματική κάρτα, αφού δεν αναγνωρίζεται το επάγγελμά μα. Επίση, οι επαγγελματίε άλλων κρατών μελών δεν μπορούν να δουν να αναγνωρίζονται τα τους στην Ισπανία λόγω ε, απώλεια νομικού πλαισίου πρέπει να σας πω ότι αυτές τα, τα επαγγέλματα IT είναι πολύ υψηλής διασυνοριακής κινητικότητας και επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια των ανθρώπων και την επιχείρησή Να μην μιλήσω για την εθνική ασφάλεια. Η ζημιά είναι τεράστια για τους Ισπανούς επαγγελματίε κυρίε και κύριοι. Και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εσεί έχετε πει ότι οι επαγγελματίε άλλων κρατών δεν μπορούν να αποτελέσουν μέρο ενό ε, συλλόγου επαγγελματικού στην Ισπανία, διότι δεν αναγνωρίζουν τα προσόντα του. Και υπάρχει τεράστια ε, διάκριση ανταγωνιστική. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Ένα επαγγελματία ε, στην, Ανταλου, στην Ανταλουσία, παραδείγματο χάρη, ε, μπορεί να χρησιμοποιήσει ε, τη μάρκα, την επαγγελματική τη Ανταλουσία, αλλά αν κάποιο δεν είναι μέλος, ε, δεν είναι δηλαδή, συμβεβλημένος, πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να το κάνει. Αυτό που είναι συμβεβλημένος μπορεί να εγγυηθεί στον πελάτη ότι έχει ένα επίσημο τίτλο. Υπάρχει ένα επίπεδο ποιότητας της υπηρεσίας υπάρχει και ένα σώμα το οποίο θα μπορέσει να, να κρίνει αν υπάρξει κάποια διαφορά. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει κάποιο που δεν είναι συμβεβλημένο. Δεν πρόκειται απλά για ε, διοικητικό ζήτημα. Πρέπει κάποιο να εγγυάται ότι πληρώνονται οι προποθέσει. Και αυτό μπορεί να το κάνει αυτό που είναι συμβεβλημένο. Αυτό που δεν, που δεν είναι συμβεβλημένο δεν μπορεί. Έχει κάλυψη σε ό,τι αφορά την παροχή των υπηρεσιών. Επίσης ε, καθορίζονται και ευθύνε για το άτομο και τι υπηρεσίε που παρέχει. Τον διέπει μια ευθύνη. Αυτό δεν ισχύει για το μη συμβιβλημένο. Επίση έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για να αναπτυχθεί επαγγελματικά. Οι τιμέ είναι πολύ χαμηλότερε για αυτόν. Επίση να υπενθυμίσω ότι οι υπηρεσίε που παρέχουμε εμεί επηρεάζουν άμεσα τη φυσική και οικονομική ασφάλεια των προσώπων και των επιχειρήσεων και σε ορισμένε περιπτώσει και το περιβάλλον αλλά και την εθνική ασφάλεια. Έτσι λοιπόν πώς μπορούμε να προστατεύσουμε την οικονομική και φυσική ασφάλεια των προσώπων, ε, η εθνική ασφάλεια, αν δεν μπορούμε να αγγιηθούμε την προσοχή υπηρεσιών και δεν ζητήσουμε να υπάρχει, δεν υπάρχει ένα πλαίσιο. Δεν να εφαρμόσουμε τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων κυβερνοασφάλεια, εφόσον το άμεσα ε, εμπλεκόμενο επάγγελμα στον τομέα αυτών δεν ρυθμίζεται. Δεν είναι θέμα αναγνώριση των προσόντων. Υπάρχει και αυτό, αλλά είναι θέμα ανταγωνιστικότητα τη ευρωπαϊκή αγορά και προστασία των καταναλωτών και των χρηστών. Επίση, πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει καμία βούληση από τι Ισπανικέ Αρχέ να επιληθεί ένα θέμα το οποίο υπάρχει εδώ και 9 χρόνια. 9 χρόνια. Αυτή τη στιγμή αναθεωρείται ε, το νομικό πλαίσιο το ευρωπαϊκό για να προσαρμοστεί στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Αναγνώριση των Δεξιοτήτων. Ωραία. Όχι όμω μένουμε εκτό αυτή τη νομοθεσία, αλλά ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει να υπάρξει αναγνώριση, ε, δεν ακούει η κυβέρνηση. Είναι σαφές στο άρθρο 36 του συντάγματος ότι ο νόμος θα καλύπτει τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων επαγγελμάτων. Αυτό λέει το Σύνταγμα το Ισπανικό. Τελειώντας να πω ότι θα πρέπει η Ισπανία να συμμορφωθεί και, αν, και θα πρέπει να επιμείνουμε να καλυφθεί και αυτό το επάγγελμα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Έχουν ήδη χαθεί 9 χρόνια κυρίε και κύριοι. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε όλο και λιγότερα μέλη στην ομάδα. Η Επιτροπή όμω είναι εδώ. Και με τα χαρά σας δώσω το λόγο για να προσπαθήσετε να εξηγήσετε την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε για το θέμα που έχει τεθεί έχουμε λάβει αναφορά από τον ίδιο τον αναφέροντα απευθείας και την εξετάζουμε εδώ και κάποιο καιρό και το ερώτημα που τίθεται είναι εάν το επάγγελμα των ε, ε, ειδικών στην πληροφορική έχει ε, ρυθμιστεί στην Ισπανία ή όχι. Από τη στιγμή που είναι ρυθμισμένο ένα επάγγελμα, εννοώ ως προς την συμπερίληψή του στην νομοθεσία, αν υπάρχει νόμος ή κανόνας που προβλέπει ότι πρέπει κάποιο να κατέχει επαγγελματικό τίτλο για να ασκήσει το επάγγελμα. Η απάντηση είναι ναι. Το επάγγελμα αυτό είναι ρυθμισμένο, άρα η Ισπανία υποχρεούται να ε, μεταφέρει την οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα και στην περίπτωση των ε, ειδικών ε, μηχανικών τεχνολογιών της πληροφορικής. Η Ισπανία δεν έχει γενικό νομοθεσία που να επιβάλλει επαγγελματικό τίτλο για ένα επαγγελματικό προσόν για την ε, άσκηση του επαγγέλματο του μηχανικού τεχνολογιών τη πληροφορική. Όμω σε διάφορε επαρχίες και περιφερειέ υπάρχουν επαγγελματικέ ε, ενώσει. Οι επαγγελματικέ αυτέ ενώσει και σύλλογοι επιβάλλουν την ε, προσχώρηση ω μέλου σε αυτήν την ένωση ή σωματείο για να μπορεί κανεί να ασχίσει το επάγγελμα. Αυτή λοιπόν στιγμή απαιτείται αυτό, απαιτείται και επαγγελματικό τίτλο. Άρα για μα η κατάσταση είναι ξεκάθαρη. Το επάγγελμα είναι ρυθμισμένο. Οι Ισπανικέ αρχέ υποχρεούνται να ε, μεταφέρουν την οδηγία. Γι' αυτό λοιπόν ήρθαμε σε επαφή με τι Ισπανικέ αρχέ για να του επιστήσουμε την προσοχή στο θέμα αυτό και μα είπαν ότι η κατάσταση εντωμεταξύ έχει αλλάξει. Δηλαδή, οι συμμετοχή, η προσχώρηση στο επαγγελματικό σωματείο δεν είναι υποχρεωτική Εκτό και αν κάποιος νόμος σε εθνικό επίπεδο επιβάλλει την προσχώρηση σε αυτό το νόμο. Για τους μηχανικούς ε, των τεχνολογιών τη πληροφορική, η προσχώρηση στο επαγγελματικό σωματείο δεν επιβάλλεται, άρα ε, δεν ε, απαιτείται για την άσκηση του επαγγέλματο και είναι τελείω εθελοντική, εθελούσια. Άρα, ένα τεχνικό ε, τεχνολογιών τη πληροφορική από άλλο κάτω μέλο μπορεί να πάει στην Ισπανία και να ασκήσει το επάγγελμα αυτό χωρί να χρειαστεί να αναζητήσει την αναγνώριση των επαγγελματικών του προσόντων δεν έχει και καμία υποχρέωση να προσχωρήσει στο επαγγελματικό σωματείο, στην επαγγελματική αυτή ένωση. Εμεί λοιπόν φροντίσαμε να κάνουμε και μια έρευνα για να δούμε στην πράξη εάν το γεγονό να μην είναι κανεί μέλο σε σωματείο ή ένωση ε, επιτρέπει να ασκήσει παρόλο το επάγγελμα όντω στην πράξη. Και αναφέρθηκε και το θέμα τη θεώρηση. Για να δούμε αν μπορεί να απαιτηθεί από τον πελάτη προκειμένου να αποδεχτεί ένα πρόγραμμα, μια πρόταση. Είδαμε λοιπόν ότι οι απαιτήσει αυτές δεν είναι τελείως υποχρεωτικέ. Οι Ισπανικέ αρχέ μάλιστα μα απήντησαν ότι αυτή η περίφημη βίζα δεν είναι ε, υποχρεωτική και ότι δεν υπάρχει μονοπόλιο. Υπάρχουν και άλλες επαγγελματικέ ε, ενώσεις ή σωματεία τα οποία μπορεί να προσχωρήσει ένας μηχανικός τεχνολογία τη πληροφορική για να ζητήσει να το επιτραπεί άσκηση των επαγγελματικών του ε, δεν έχουμε λάβει κανένα παράπονο από μηχανικό τεχνολογιών τη πληροφορική από άλλο μέλο που παραπονέθηκε ότι δυσκολεύεται να ασκήσει το επάγγελμα του στην Ισπανία. Σε αυτή τη φάση λοιπόν δεν υπάρχει κανένα φραγμό για να ασκηθεί το επάγγελμα αυτό στην Ισπανική αγορά και προφανώ η, η Ισπανία δεν χρειάζεται και να μεταφέρει την οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητε, διότι δεν χρειάζεται να πετυχθεί η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων προηγουμένω για να ασκηθεί το επαγγέλμα αυτό. Σε ό,τι αφορά του μηχανικού από την Ισπανία που θα ήθελαν να ασκήσουν την επαγγελματική του δραστηριότητα σε ένα άλλο κράτο μέλο, η οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητε εφαρμόζεται πλήρω. Απλώ τα άλλα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα, όπω το επαγγελματέ ρυθμίζεται στην Ισπανία, να απαιτήσουν απόδειξη επαγγελματική πείρα ενό τουλάχιστον έτου σε ένα κράτο μέλο που δεν ρυθμίζει το επάγγελμα αυτό προτού εφαρμόσουν τα τη οδηγία. Πάντω, ακόμα και αν η οδηγία δεν ισχύει, τα άλλα μέλη που θα λάβουν αιτήματα αναγνώριση ε, από μηχανικού τη Ισπανία έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν τη συνθήκη. Δηλαδή, ακόμη και αν δεν εφαρμόζεται η οδηγία, δεν σημαίνει ότι για την επαγγελματική πιστοποίηση δεν υπάρχουν κανόνε που έχουν επιβληθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το θέμα αυτό. Να προσθέσω ότι ουδέποτε λάβαμε προσφυγή παράπονο ή αναφορά από μηχανικό τεχνολογιών πληροφορικής από την Ισπανία που να αναφέρει δυσκολία να ασκήσει το επαγγελμά του σε άλλο κάτω Η δική μα λοιπόν πρόθεση από τη δική μα την υπηρεσία είναι να ζητήσουμε να κλείσει η εξέταση αυτή τη αναφορά. Έχουμε ετοιμάσει σχετική επιστολή τη ε, αρχική ε, τήρηση στα αρχεία τη αναφορά αυτή προ τον αναφέροντα Εκτό και αν μα παρουσιάσει κάποια σαφή απόδειξη ότι υπάρχει μια κατάφορη παραβίαση των κανόνων, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία τέτοια απόδειξη. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε εμεί. Ο λόγο στου συναδέλφου, εφόσον τον επιθυμούν. Πέτερ. Με μπέρδεψαν κάπω αυτά που άκουσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχάς, ε, εντάξει, στην αρχή μου φάνηκε λογικό αυτό που είπε η Επιτροπή, ότι η Ισπανία ασκεί τα δικαιώματά της, ο αναφέρον όμως έχει διαφορετική άποψη. Και πρέπει να πω ότι πάντα τη στιγμή που λέω «Α, εντάξει, κατάλαβα τι γίνεται», τότε ε, καταλαβαίνω ότι δεν ξέρω τίποτα. Νομίζω πως ε, για μένα το βασικό ερώτημα είναι τα δικαιώματα που έχει ένας τεχνικός μηχανικός πολεμιστών στην Ισπανία ε, και αυτά που έχει ένας ε, άλλος, ένας υπήκος άλλου κράτους μέλους. Και, και επίσης ε, πρέπει να δούμε τη διαφορά ανάμεσα σε έναν αλλοδόπο που εργάζεται, που θέλει να εργαστεί στην Ισπανία και σε έναν Ισπανό που θέλει να εργαστεί στο εξωτερικό. Εδώ πράγματι υπάρχουν διαφορές, αλλά το θέμα είναι αν γίνονται διακρίσεις από την ισπανική πλευρά. Και η Κομισιόν μας λέει ότι η Ισπανία έχει δικού της νόμους, έχει ρυθμίσει με δικό της ε, τρόπο το θέμα και αυτό μπερδεύει τα πράγματα. Όταν κάποιος, ας πούμε, έχει σπουδάσει στη Γαλλία, υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, αναγνώριση στοιχείου κτλ. Κάποιες διαδικασίες ε, αναγνώρισης. Αυτό όμως με μπέρδεψε, δεν, ομολογώ πως δεν το κατάλαβα. Ο αναφέρον μας λέει πως υπάρχει πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Όσοι συνάδελφοι έχουν μείνει νομίζω πως ε, δεν είναι σε πολύ καλύτερη θέση από μένα. Αλλά ίσως εκείνοι ξέρουν, έχουν μια πρόταση για το πώς να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, Άντζελα. Εγώ γνωρίζω Το πρόγραμμα το πρόβλημα αυτό. Ξέρω ότι οι άνθρωποι αυτοί ε, δεν μπορούν να εργαστούν. Εδώ και το, το πάρκμα της Γερμανίας. Εδώ δεν σεβόμαστε ένα βασικό δικαίωμα. Έτσι λοιπόν εγώ θα ζητούσα να παραμείνει ανοιχτό το θέμα. Εάν χρειαστεί να φέρει περισσότερα στοιχεία αναφέρον, να, να το συμπληρώσει, να μας τα διαβιβάσει, να τα στείλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να υπάρξει μια ενημέρωση για το θέμα αυτό, αυστηρά, να απευθυνθεί ξανά στι Ισπανικές Αρχές ενδεχομένω, με τις νέες πληροφορίε που θα δώσει ο αναφέρον. Ε, να μα εξηγήσουν δηλαδή οι Ισπανικές Αρχές τελικά τι συμβαίνει. Διότι οι επιπτώσει είναι σαφές. Λέτε εδώ ότι όλα είναι καλά, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μάλιστα. Μπορούμε να δώσουμε τώρα το λόγο στον αναφέροντα. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ναι, για να απαντήσω στα, στο μέλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι μόνο υπάρχουν προβλήματα να εργαστεί κάποιο να παρέχει υπηρεσίε εκτό τη Ισπανία, είναι ότι δεν μπορεί να παρέχει κάποιε υπηρεσίε ούτε στην ίδια την Ισπανία, που είναι και το χειρότερο. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Εγώ να σα πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, το δικό μου. Εγώ είμαι υπεύθυνο πληροφορική στον τομέα δικαστικό. Ε, ε, μπλέκομαι στα δικαστήρια δηλαδή. Και εδώ συμμετέχουν κάποιοι οι οποίοι ε, έχουν πτυχία, κάνουν αυτή τη δουλειά και έχουν πτυχία καλών τεχνών. Τι σχέση και αυτό με την πληροφορική, τίποτα. Ε, δεν υπάρχει σύμβαση συλλογική ε, για τον τομέα των TIC, των νέων, τεχνολογιών δηλαδή, ενώ θεωρείται ότι αυτό επηρεάζει άμεσα την εθνική ασφάλεια. Εμένα μου φαίνεται απίστευτο. Είναι κάτι που επηρεάζει άμεσα την εθνική ασφάλεια και δεν ρυθμίζεται η παροχή υπηρεσιών. Θα πάρουμε δηλαδή, θα, θα, να απελευθερώσουμε και τι υπηρεσίε τη ιατρική, τα πάντα, να κάνει ο καθένα ό,τι θέλει. Δεν το αντιλαμβάνομαι, δεν το καταλαβαίνω. Είναι αυτό που σα λέω. Δεν μπορούμε να ασκήσουμε το ίδιο το επάγγελμά μα στην Ισπανία, στη χώρα μα. Δεν σας λέω έξω, από την Ισπανία. Στην ίδια την Ισπανία. Εγώ έχω μια, ε, μια επιστολή που μου έστειλε ε, η υπηρεσία απασχόληση τη χώρα μου που λέει ότι επειδή εγώ δεν έχω κάνει ένα μάθημα 30 ωρών ότι μπορώ, ότι, ότι ξέρω να χρησιμοποιήσω έναν ε, ε υπολογιστή ε, ενώ έχω δίπλωμα ε, ειδικού πληροφορική μου λένε ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν υπολογιστή. Ε, από το 2009 είναι έτσι τα πράγματα και έχουμε πραγματικά φτάσει στα όρια μα. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Η Ισπανία είναι λίγο μακριά από τι Βρυξέλλε, αλλά το πρόβλημα αυτό είναι ένα χοντρό πρόβλημα. Ε, και εδώ από το 2008 ε, πιέζουμε γι' αυτό. Το ίδιο το Ισπανικό Σύνταγμα λέει ότι πρέπει να ρυθμίζεται η άσκηση ενό επαγγελματο από νόμο. Δεν είμαστε λοιπόν ε, επάγγελμα το οποίο έχει ένα συγκεκριμένο τίτλο. Είμαστε. Δεν μπορεί κανεί να το αμφισβητήσει αυτό. Φέρνουμε στοιχεία εδώ και τρία-τέσσερα χρόνια. Και μπορούμε να φέρουμε και άλλα στοιχεία. Αλλά αυτό που θέλουμε είναι λύσει κάποια στιγμή. I think I saw that you wanted to come in again. Can you do that very, very briefly? Ναι, καταλαβαίνω ότι το πρόβλημά σα αφορά το εσωτερικό τη Ισπανία όμω. Εδώ δεν είμαστε ο κατάλληλο συνομιλητή, διότι αν μηχανικοί με προσόντα στην Ισπανία έχουν δυσκολίε να βρουν δουλειά στην Ισπανία, αυτό αφορά την Ισπανία. Νομίζω ότι αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θέλετε η Ισπανία να αναλάβει τη ρύθμιση του επαγγέλματο. Εδώ και πάλι δεν είμαστε εμεί ο κατάλληλο συνομιλητή. Ο δικό μα στόχο δεν είναι να πιέσουμε τα κατημέλη να γκρίνουν νομοθεσία. Ε, σα ίσα. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια ανεβαία αναγνώριση των ρυθμισμένων επαγγελμάτων που καλύπτουν όλα τα επαγγελμάτα και όλου του επαγγελματικού κλάδου όλα τα κατημέλη και καλέσαμε να εξετάσουν όλου του κανόνε του για να δουν αν είναι δικαιολογημένοι ή όχι. Ο στόχος λοιπόν προφανώς δεν είναι να αρχίσουμε να πιέζουμε να υπάρχει απορρίθμιση, διότι προφανώς χρειάζονται κανόνες. Όμως καταλαβαίνετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να πιέσει ένα κάτω μέλος να προβλέψει κάτι και να δημιουργήσει φραγμό στην ελεύθερη κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά. Δεν είναι κάτι το καινούριο. Διαρκώς δεχόμαστε ε, κλήσει από, ευρωπαϊκά, από επαγγελματικά σωματεία, επαγγελματικέ ενώσει που έρχονται να μα μιλήσουν για να πιέσουμε να υπάρξει ρύθμιση, να πιέσουμε να αυξηθούν οι απαιτήσει. Δεν είμαστε όμω ο κατάλληλο συνομιλητή, λυπούμε. Δικό μα προτεραιότητα είναι να δημιουργήσουμε μια μεγάλη εσωτερική αγορά χωρί φραγμού. Δεν είμαστε ε, καουμπόιδες κατά της οποιασδήποτε βέβαια ρύθμισης και του οποιοδήποτε κανόνος όμως εάν οι Ισπανικές αρχές δεν το επιθυμούν εμείς δεν μπορούμε να τις υποχρεώσουμε ούτε να τις πιέσουμε να προβλέψουν ε, κανόνες δεν έχουμε δυστυχώς τις ίδιες προθέσεις Σας ευχαριστώ πολύ Πέτερ Εγώ όμως έχω εξακολουθώ να έχω ένα αναπάντητο ερώτημα τι ακριβώς γίνεται στην περίπτωση της Ισπανίας Στη Γερμανία όταν προκυρήσεται διαγωνισμός για μία θέση τότε αναφέρονται ε, με κάθε λεπτομέρεια τα προσόντα που χρειάζονται ε, και δεν μπορεί κανείς να ε, πει ότι εδώ πέρα γίνονται διακρίσεις ή οτιδήποτε. Όταν θέλω κάποιον πληροφορικάριο θέλω έναν που να έχει αυτό και αυτό και αυτό το προσόν. Και πάλι εξακολουθώ να είμαι μπερδεμένο με την απάντηση της Κομισιόν. Εντάξει, στην Ισπανία έχει δίκιο βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορούμε να ανακατευτούμε στα δικά τους ε, χωράφια, αλλά μου φαίνεται πως υπάρχει εδώ διάκριση, διότι οι Ισπανοί τεχνικοί μηχανικοί πληροφορικοί δεν μπορούν να εργαστούν στο εξωτερικό. Αλλά εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει πως δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα, μήπως επειδή δεν έχουν έτσι κι αλλιώς καμία ελπίδα. Εντάξει, όταν είσαι πληροφορικάριος έχεις επιλέξει ένα επάγγελμα με υψηλές απαιτήσει. Όποια θέση και να ζητήσεις, σε οποιαδήποτε επιχείρηση, πάντα θα υπάρχει θέση για έναν πληροφορικάριο. Θα έπρεπε λοιπόν να είναι εύκολο κάποιος να βρει δουλειά οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να αναγνωρίζετε τα προσόντα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βαλίνα, θέλετε κι εσείς να τοποθετηθείτε. Ναι, πολύ σύντομα. Συμφωνώ απόλυτα με τον Πίτερ και διαφωνώ απόλυτα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ ότι αν κάποιο δεν μπορεί να εργαστεί σε άλλο κράτο μέλο, όχι μόνο ε, στην δική του, αλλά σε άλλε χώρε, δεν υπάρχει πρόβλημα ελεύθερη κυκλοφορία. Ε, και βεβαίω και επηρεάζει. Είναι λοιπόν απαραίτητο να το διευκρινίσουμε αυτό να το αφήσουμε ανοιχτό και να συλλέξουμε όλες τις πληροφορίες που πρέπει να συλλέξουμε. Okay, let's... Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ας το κάνουμε λοιπόν αυτό. Ας αφήσουμε την αναφορά ανοιχτή και μπορούμε να απευθυνθούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περαιτέρω πληροφορίες. Νομίζω πως κάνατε ό,τι μπορούσατε βέβαια αλλά αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να στείλουμε μία επιστολή που θα εκφράζει τις ανησυχίες μας για την κατάσταση στην Ισπανία. Και επίσης να φροντίσουμε έτσι ώστε ο αναφέρον να στείλει περισσότερες πληροφορίες και να είμαστε σίγουροι πως έχουμε διερευνήσει την κάθε λεπτομέρεια προτού κλείσουμε την αναφορά. Έτσι λοιπόν θα πράξουμε. Και τώρα 6 και 18 ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι καλό βράδυ και ε, σας εύχομαι καλή τύχη, καλή επιστροφή στην Ισπανία κύριε και απολαύστε τη λιακάδα των Βρυξελών.